First of all, I want to... Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς να δώσω το λόγο στους διερμηνείς ε, που συνεχίζουν την σκηνητοποίησή ε, τους. Ε, σας ζητώ λοιπόν να φορέσετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τη δήλωσή τους. Παρακαλώ, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στους διερμηνείς. Καλημέρα σας. Ε, βρισκόμαστε στην 24η μέρα των κινητοποιήσεών μας και ακόμα δεν έχουμε δει καμιά θετική αντίδραση εκ μέρους της διοίκησης. Αντίθετα, ο Γενικός Γραμματέας κληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του. Στη σημερινή συνεδρίαση, πολλοί συναδελφοί μας από άλλες καμπίνες έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Σε ένδειξη αλληλεγγύης, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασίας όπως αρχικά προβλεπόταν, ωστόσο η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώς στην προγραμματισμένη ώρα λήξη της Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή προσοχή η Πρόεδρος. Και τώρα, ω ήθιστε, πρώτο σημείο είναι η, μερίσια, η έγκριση μάλλον τη ημερήσια διάταξη. Πρέπει να, να βάλουμε την ψηφοφορία για την υπόθεση των ανανεώσιμων, γιατί υπάρχουν κάποια μικρά ζητήματα που πρέπει να αποσαφενιστούν ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο μετά από την χτεσινή σύσκεψη. Ε, δεν υπάρχουν αντιρρήσει, λοιπόν, να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη με αυτήν την αλλαγή. Ωραία, λοιπόν. Οπότε, έχω να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Στην συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου, οι συντονιστές αποφάσισαν να εφαρμόσουν την διαδικασία του ε, κανονισμού 53 4 ε, που ε, καθορίζει την μορφή της τροπολογίας για τον φάκελο αυτό, για το θέμα αυτό τα βενθοπελαγικά είδη στην Δυτική Μεσόγειο, πολιετές σχέδιο. Εδώ λοιπόν ε, είπαμε ότι θα κάνουμε μία τοποθέτηση υπό τη μορφή ε, τροπολογιών. Δεν έχουμε λοιπόν ε, συντάκτη γνωμοδότηση, δεν θα κάνουμε γνωμοδότηση. Θα δούμε λοιπόν, τις, ε, θα υποβάλουμε τις απόψεις μας άμεσα στην ε, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, στην Επιτροπή Αλληλείας ε, υπό τη μορφή τροπολογιών. Η, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην ΕΝΒΗ είναι η 5η Ιουλίου στις 11 και η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ θα προγραμματίζεται για τις 13 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Επίσης, εν ώψη του μεγάλου φόρτου εργασίας προς το τέλος της θητείας, οι συντονιστές αποφάσισαν να αφήσουν την, να ανοίξουν την προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για διάφορα θέματα. Οπότε δεν έχουμε ε, συντάκτη γνωμοδότηση στην ΕΜΒΗ και δεν θα υπάρξει σχέδιο γνωμοδότηση. Σας θα σας πω τους φακέλους που δεν θα κάνουμε γνωμοδοτήσεις. Θα υιοθετηθούν εδώ λοιπόν οι τροπολογίες και θα θεωρηθούν ως γνωμοδότηση ε, δική μου του Πρόεδρου. Αυτό έχει να κάνει με τη συμπλήρωση της ε, έγκρισης τύπου ε, σε σχέση με την απόσταση του Ηνωμένου Βασιλείου από, το, από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προθεσμία είναι 5η Ιουλίου. Ε, και θα ψηφιστεί 29-30 Αυγούστου. Μετά έχουμε το SEF, Connecting Europe Facility, η προθεσμία είναι 11 Ιουλίου και η ψηφοφορία είναι 10 με 13 Σεπτεμβρίου. Μετά αποκάλυψη σχετιζόμενη με βιώσιμες επενδύσεις και βιώσιμους κινδύνους. 4 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία και ψηφίσουμε τον Οκτώβριο. Και επίσης και κανονισμός περί κοινών διατάξεων Έχουμε προθεσμία υποβολής τροπολογιών στην ΕΝΒΗ 5 Σεπτεμβρίου και η ψηφοφορία θα γίνει τον Οκτώβριο. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και ως ήθιστε έχετε λάβει τους φακέλους σας ηλεκτρονικά και η συνεδρίασή μας αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Ε, τώρα έχουμε σύσταση των συντονιστών από τις 21 Ιουνίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Το ίδιο ισχύει για τα πρακτικά της συνεδρίασής μας από τις 19 και 20 Μαρτίου και από τις 26-27 Μαρτίου. Θεωρούμε πως εγκρίνονται εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Τώρα, συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Περί των κανόνων για τη διάθεση στην αγορά ε, Κατά τον τρίτο τριμερή που έγινε στις 19 Ιουνίου αρκετά, συζητήθηκαν αρκετά πολιτικά και τεχνικά θέματα ε, συμπεριλαμβανομένων των ε, ορίων Καδμίου, όπου έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Στο τέλος του τριμερού, στο Συμβούλιο κατέστησε σαφές ότι είναι πρόθυμο να κάνει υποχωρήσεις προς το Κοινοβούλιο για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, εφόσον το Κοινοβούλιο δεχτεί τον ορισμό ε, ορίου για το κάδμιο 60 mg ανά κιλό και να μην μειώσει άλλο το, αυτό το, όριο. Όμως το Κοινοβούλιο διατήρησε τη θέση του για τα όρια περί καδμίου και δεν επετέφθη συμφωνία. Από ό,τι εγώ ο το θέμα θα πάει και θα περάσει στην Αυστριακή Προεδρία. Πρόωθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναθεώρηση Recast. Επετέθη συμφωνία στον πέμπτο τριμερή που έγινε στις 13 Ιουνίου. Συμφωνήσαμε προσωρινά για ένα μέρος ενέργειας από ανανεώσιμες, της τουλάχιστον 32% ε, μέχρι το 2030 όσον αφορά την μεχτή τελική κατανάλωση της Ένωσης με ανωδική ε, ρήτρα αναθεώρησης με το 2023. Επίσης συμφωνήθηκε ένα μήνυμο μερίδιο του 14% που για τις μεταφορές που πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Ιδιαίτερα τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς που βασίζονται σε ε, καλλιέργειες ε, τροφίμων θα πρέπει να φτάσουν στο ανώτατο όριο του 2020 με ένα έξτρα 1% και σε καμία περίπτωση να μην ξεπεραστεί το 7% για την τελική κατανάλωση στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Και το μερίδιο των προηγμένων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου ε, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1% το 2025 και 3,5% στο 2030. Ε, επίσης, ε, τα βιοκάψιμα από καλλιέργειες τροφίμων όπως ε, το φινικέλαιο, τα τα οποία έχουν επιπτώσεις στην χρήση γης θα πάψουν να χρησιμοποιούνται σταδιακά μέσω μιας διαδικασίας πιστοποίησης η οποία θα συσταθεί. Θα ψηφίσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, μάλλον τα τμήματα που αφορούν αποκλειστικά την ΕΝΒΗ θα ψηφιστούν σήμερα και στην Ήτρη η ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουλίου. Η ψηφοφορία στην Ήτρε 10 Ιουλίου, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, η διακυβέρνηση στην ε, Ενεργειακή Ένωση. Έχουμε φτάσει σε μια προσωρινή συμφωνία στις 19 Ιουνίου οι δύο συνομοθέτες συμφώνησαν για βασικά πολιτικά θέματα σε μια δέσμη που περιλαμβάνει μια σταθερή, ένα σταθερό και ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τα κράτη-μέλη. Καλύπτουν όλες οι διαστάσει τη Ενεργειακή Ένωση και λαμβάνονται υπόψη η μακροπρόθεσμη προοπτική. Μια μακροπρόθεσμη στρατηγική περιλαμβάνει μια ανάλυση που καλύπτει το σενάριο επίτευξη ε, για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών του αερίων του θερμοκηπίου μέχρι ε, το, το 2050 στην Ένωση. Ο ορισμός ε, ε, της αρχής για την απόδοση της ενέργειας πρώτα απ' όλα, ή διατάξεις για την εξασφάλιση της συνέχειας που θα δοθεί στους, στην πρόοδο που, που σημειώνουν τα κρατημέλη Επίσης ε, ε, θεσπίστηκε ο στόχος για τα ανανεώσιμες. Όλα αυτά έγιναν δεκτά από το Συμβούλιο και έτσι φτάσαμε σε συμφωνία. Τώρα, ορισμός παρουσίαση και ετικετοθεσία των αλκοολούχων ε, ποτών. Στον δεύτερο άτυπο τριμερή που έγινε στις 27 Ιουνίου, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν είχαν μια παραγωγική ανταλλαγή απόψεων που καλύπτουν τις ε, βασικές πτυχές των θέσεών τους. Η συζήτηση ήδη έθιξε πολλά ζητήματα που σχετίστηκαν με τη μεταβατική περίοδο ε, όπως ας πούμε γεωγραφικές ενδείξεις και οι σχετικοί ορισμοί. Υπάρχει η δυνατότητα συμφωνίας. Ωστόσο, δεδομένης ε, της ε, ε, μεγαλύτερης, μάλλον υπεροχής των τεχνικών θεμάτων που εξετάζονται σε αυτή την πρόταση, η Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν να, να, να, παραπέμψουν σε τεχνικό επίπεδο την προετοιμασία του μελλοντικού τριλόγου, τριμερούς δηλαδή διαλόγου, που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Τώρα, Πάμε στο πρώτο σημείο της σημερινής μας ε, διάταξης, ε, τη χρήση της κανάβεως για θεραπευτικούς σκοπούς. Έχουμε διάφορους εισηγητές. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο από το ΕΛΚ είναι η κυρία Σουίτσα. Α, δεν είναι εδώ. Έπειτα έχουμε τους σοσιαλιστές, τον κύριο Μπαλάς. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλετε να αρχίσω αμέσως. Πολύ ωραία. Δεν το συνηθίζω, αλλά θα σας διηγηθώ κάτι που μου συνέβη πριν από λίγα χρόνια, όπου ασθένησα από την αρρώστια του Λάιμ με πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Είχα πολλούς, πολύ έντονους πόνους και είχα πάει σε ένα Γάλλο γιατρό. Τότε όλες οι μορφές κανάβες ήταν πρόσθετες και απαγορευμένες. Οπότε ο γιατρός μου είπε ε, έχουμε, και μάλιστα ένας κορυφαίος γιατρός, είπε η μόνη λύση για να καταπραϊνθούν οι πόνοι σας είναι να χρησιμοποιήσετε κάναβη. Εγώ είπα όμως δεν θέλω να καταστρατηγήσω την νομοθεσία της χώρας. Υπάρχει ε, πρόσβαση σε νόμιμες μορφές κάναβης. Μου είπε όχι σήμερα δεν επιτρέπονται ακόμη. Υπάρχει όμως μου είπε ο γιατρός αυτός ότι δύο είναι οι δραστικές ουσίες ε, της κάναβης. Ένα συστατικό είναι ψυχοτρόπο Οπότε αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε γιατί είναι πολύ ε, επιζήμιο και προκαλεί φοβερές βλάβες. Αλλά υπάρχει και άλλη δραστική ουσία στην κάναβη που είναι χαλαρωτική, έχει χαλαρωτική επίδραση και μπορεί να καταπραίνει τους πόνους. Γνωρίζουμε τώρα ότι και από επιστημονική άποψη υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό των δύο δραστικών συστατικών. Μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε την καναβιδιόλη, το CPD, για τι χημειοθεραπείε, ε, στη θεραπεία του καρκίνου δηλαδή, Επίσης μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για την ασθένεια του κρόνου, για τη σκλήριση κατά πλάκας, για την ασθένεια του λάιμ και για τη σκλήριση κατά πλάκας όπως είπα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στους ασθενείς σε αυτή τη δραστική ουσία, την καναβιδιόλη, ώστε να έχουν μείωση των πόνων τους, το ελάχιστο. Βέβαια δεν έχουμε εναρμονισμένη νομοθεσία στα κράτη-μέλη όπως θα φαντάζεστε για το θέμα αυτό. Οπότε δημιουργείται πολύ άνηση πρόσβαση στα προϊόντα αυτά για του ασθενεί. Δεύτερο πρόβλημα, δεν έχουμε κατά ανάγκη ασφαλή προϊόντα. Αυτό είναι ένα άλλο μείζον ζήτημα. Μερικέ φορέ έχουμε κακή ποιότητα προϊόντα που δεν ανταποκρίνονται στα ιατρικά κριτήρια και στι προδιαγραφέ και αυτά κυκλοφορούν στην αγορά. Γι' αυτό και ζητούμε μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για την κάναβη ιατρική χρήση. Ε, θέλουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση τη έρευνα για τέτοια προϊόντα, για να γνωρίζουμε με ασφάλεια και βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τη χρήση τέτοια ε, δραστική ουσία, τη CBD, τη καναβιδιόλη δηλαδή, στην κάναβη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το επισημάνουμε και να δούμε τι αλληλεπίδραση έχει αυτή η δραστική ουσία με άλλες ε, δραστικές ουσίες ότι θετικές επιδράσει αρνητικές ενδεχομένω. ώστε να έχουμε μια σαφή γνώση της κατάστασης. Θέλουμε πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα για τους ασθενείς και να επιτρέψουμε στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, γιατί μέχρι στιγμής η καινοτομία για τέτοια προϊόντα προέρχεται από τρίτες χώρες. Μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να βάλουμε τον ασθενή στο επίκεντρο της ε, πολιτικής. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε καλύτερη κατάρτιση των επαγγελματιών τη υγεία, για να μπορούν καλύτερα να συμβουλεύουν και να παραστέκονται στου ασθένειε κατά τη διάρκεια τη ε, θεραπευτική αγωγή. Επίση, ε, και η φαρμακοποίηση θα πρέπει να ενημερώνουν. Τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι ένα τμήμα τη λύση. Γιατί να μην έχουμε και φυτοθεραπευτικά προϊόντα με βάση την ε, φαρμακευτική κάναβη. Και θα πρέπει να γίνει μια στάθμιση των δραστικών ουσιών. Ή επίση ε, να έχουμε οριοθετημένη την καλλιέργεια στο σπίτι για κατανάλωση. Θα πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε στου ασθενεί που υποφέρουν από χρόνιους πόνου την καλύτερη δυνατή προστασία και γι' αυτό κρίνουμε το ψήφισμα αυτό σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Κρούπα. Ευχαριστώ. Όντως, το σχέδιο ψηφίσματος ε, στη μορφή που έχει αξίζει συζήτησης και επεξεργασίας. Γιατί επικρατεί τεράστιο χάος στην νομοθεσία για την ε, ε ιατρική μαριχουάνα. Γιατί δεν έχουμε μόνο δύο δραστικές ουσίες ε, στην κάναβη. Έχουμε περίπου 500 ενώσεις στην κάναβη και συνεχώς ανακαλύπτονται καινούριε. Οπότε το θέμα της επεξεργασίας τέτοιων προϊόντων είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται κάποια απομόνωση συγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Εγώ για 40 χρόνια ήμουν γιατρός και πρώτη φορά συνάντησα τέτοια διάσταση απόψεων για, μια συγκεκριμένη, για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Και μάλιστα ακόμη ολόκληροι καθηγητές με τίτλους και πτυχία έχουν διαφορετική άποψη μερικοί είναι υπέρ της χρήσης για κάποιους ε, σκοπούς, ε, για, για χρόνιους πόνους και κάποιες ασθένειες, αλλά υπάρχει και η αντίθετη επικριτική άποψη εις βάρος της χρήσης της ιατρικής κάναβης. Θα πρέπει λοιπόν ε, να χρηματοδοτήσουμε ανεξάρτητες μελέτες για την μελέτη αυτών για την εξέταση αυτών των προϊόντων. Γιατί υπάρχει τεράστιο χάος από μεροληπτικές μελέτες που χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ από την ιατρική βιβλιογραφία γνωρίζω για πολλές παρενέργειες ε, αλλά και για θετικές ενέργειες καναβιδιόλης ε, σε σπαστικότητα που προκαλούν κάποιες νόσες. Ούτε και γι' αυτό υπάρχουν αρκετά ιατρικά στοιχεία. Ε, γιατί αναφέρεται ότι βοηθά τη σπαστικότητα η καναβιδιόλη, αλλά δεν είναι αποδεδειγμένο πάντα. Επίσης, έχουμε πάρα πολλά παυσίπονα, όχι μόνο πιούχα που είναι παυσίπονα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εκπονήσουμε εμπεριστατωμένες μελέτες και κυρίως να ζητήσουμε ανεξάρτητες μελέτες, γι' αυτό στηρίζω και το ψήφισμα, και να διευκρινιστούν όχι μόνο αυτές οι δύο δραστικές ουσίες που αναφέρονται THS και CBD, αλλά και οι πολυάριθμες άλλες ενώσεις και θα πρέπει να αποφευθεί το εμπόριο τέτοιων ουσιών. Γιατί το Ινστιτούτο Φαρμάκων στην Πολωνία ε, είχε καλλιέργεια κάναβης και παρήγαγε το ίδιο το Ινστιτούτο Φαρμάκων Κάναβη στην Πολωνία και παρασκεύαζε τέτοια φάρμακα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Όντως χρειάζονται ε, μέσα και διεξαγωγή ανεξάρτητων αντικειμενικών μελετών. Ευχαριστώ κύριε Μπέρτερ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως ακούσαμε υπάρχουν σοβαρά επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν που λένε ότι η ιατρική κάναβη μπορεί να δώσει να έχει ανακουφιστικό χαρακτήρα για τον χρόνιο πόνο και ακούσαμε και μαρτυρία του συναδέλφου. Υπάρχει μόνο ένα φάρμακο ονόματι Savitex για την σκλήρηση κατά πλάκας που υπάρχει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγεται μάλιστα σε, από μια εταιρεία στην περιφέρειά μου. Το Savitex αυτό έχει έγκριση βάσει της αμοιβαίας αναγνώρισης, όμως της είπα θα ανακοινώσουν προσεχώς ε, ένα φάρμακο με βάση την κάναβη για την θεραπεία των συμπτωμάτων της επιληψίας και πρέπει ακριβώς ε, να υπάρχει δυνατότητα για τους ασθενείς που τα χρειάζονται. Είναι μια πραγματική ευκαιρία νομίζω. Ε, ευκαιρία αυτή την συζήτηση και την προφορική ερώτηση να συζητήσουμε λίγο με βάση την κοινή λογική και νομίζω ότι και εν ώψη των ευρωεκλογών έχουμε καθήκον να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα λογικά και ανοιχτά. Υπάρχει σύγχυση. Και εμείς στο Κοινοβούλιο αυτό γνωρίζουμε πως η διατύπωση έχει σημασία και έχει σημασία το πώς ονομάζουμε τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή λέμε καναβι. Ε, υπάρχει σύγχυση με το θέμα του παράνομου ναρκωτικού. Ίσως θα έπρεπε να μιλάμε για καναβινοειδή ή παράγωγα τετράιδρο καναβινόλης κτλ. Τα φυτικά υπάρχουν παντού στα φάρμακα. Δεν ξέρω δηλαδή αν κάποιος σήμερα ανακάλυπτε την ασπιρίνη, αν θα λέγαμε πως πρέπει όντως ε, να τα παίρνουμε από το φλοιό της ιτιάς ε, κτλ. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για την, δεν μιλάμε για την χρήση αναψυχής αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Έχουμε μια φρικτή κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα παιδάκι που η μάνα του του έδινε έλαιο κάναβης γιατί είχε πολύ σοβαρές επιληπτικές κρίσεις ε, και το κατέσχεσαν το μπουκαλάκι αυτό γιατί το θεωρούσαν κάναβη. Ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να μιλήσουμε λοιπόν για φάρμακα που προέρχονται από την κάναβη, να τα λέμε καναβινοειδή ή με το όνομα της δραστικής ουσίας για να μπουν στην αγορά και να έχουν οι ασθενείς ακριβώς ε, την ε, ανακούφιση που χρειάζονται. από Χρειάζεται λοιπόν επένδυση, χρειάζεται έρευνα κατά προτεραιότητα. Είναι πολύ φθηνό ως φάρμακο εάν εγκριθεί. Αλλά βεβαίως πρέπει να εκπαιδευτούν ε, και τα ιατρικά επαγγέλματα για την χρήση αυτών των φάρμακων. Δεν έχει νόημα δηλαδή να δώσουμε ένα φάρμακο στην αγορά χωρίς να υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση και να διαχωριστεί. Ε, δεν μιλάμε για αναψυχή εδώ πέρα, μιλάμε για ένα φάρμακο που πρέπει να δοκιμαστεί και να διατεθεί. Σα ευχαριστώ, Χάουσλινγκ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους την συνεργασία στο θέμα και συμφωνούμε σε πολλά θέματα. Πράγματι με τη χρήση καναβέως μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς ασθενείς με χρόνιους πόνους. Αυτό είναι γνωστό. Στην Ευρώπη ακόμα δεν έχουμε κάποια φάρμακα με βάση την κάναβη ε, που να έχουν αδειοδοτηθεί και θα πρέπει να φροντίσουμε γρήγορα να υπάρξει αδειοδότηση αυτών των φαρμάκων. Επίσης συμφωνώ ότι υπάρχει ανάγκη έρευνας και ότι πρέπει να στηριχθεί να καταλήξουμε σε κάποια αποτέλεσματα τα οποία θα δείξουν πόσο σημαντική θα είναι τελικά η αδειοδότηση. Υπάρχουν πολλοί λομπίστες βεβαίως ε, ε, που περιφέρονται στους διαδρόμους και προσφέρουν την δική τους ε, τετράιδρο Και ακριβώ υπάρχει αυτό το θέμα της φαρμακευτικής και ψυχαγωγικής χρήσης, δηλαδή πώς θα υπάρχει ακριβώς το θέμα του να μην ε, ε, υπάρξει διακριτική μεταχείριση της ιατρικής ε, καναβίως. Και βεβαίως να υπάρχει και η δυνατότητα ατομικής δοσολογίας. Δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το αφήσουμε στις φαρμακευτικές εταιρείες. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες επίσης για τις πρώτες ύλες και βέβαιω ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και χρόνια στη Γερμανία είναι πρόβλημα προσφοράς και έχουμε προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά. Α, δεν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό, μπορούμε να έχουμε τοπική παραγωγή. Μετά είναι επίσης σημαντικό να δούμε το θέμα της προσβασιμότητας των προϊόντων αυτών. Θεωρώ ότι εδώ πέρα έχουμε έναν αγώνα με τα ταμεία υγείας, αν θα πληρώσουν τελικά κάτι τέτοιο. Αν γίνει αυτό το βήμα και το επιτρέψουμε στην Ευρώπη και εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι είναι λογικό κάτι τέτοιο, πρέπει να φροντίσουμε και τα ταμεία υγείας να καλύπτουν τα προϊόντα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τόρες Μαρτίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όντως, στη συζήτηση αυτή μας έχει προλάβει η κοινωνία. Εμείς υστερούμε. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να αποδώσουμε δικαιοσύνη, γιατί περί αυτού πρόκειται. Να δώσουμε δικαιοσύνη, να αποδώσουμε δικαιοσύνη στους ασθενείς ε, που παραπονιούνται με το στίγμα που τους ε, έχουν κολλήσει μερικοί επειδή χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τέτοια ε, φάρμακα για να ανακουφίσουν τους πόνους τους. Η κάναβης, όπως είπαν ε, οι συνάδελφοι, έχουν, έχει αναγνωρισμένα θετικά αποτελέσματα για πολλές ασθένειες. Οπότε είναι ανήκουστο που παρά την χρήση για νόσο από AIDS, Alzheimer, αρθρίτιδα, ε, ασθένεια του Κρόνου, σκλήρηση κατά πλάκας, ε, η άσθμα. Απαγορεύεται ακόμη η χρήση για ιατρικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τι ε, να μιλούμε τόσο πολύ για την κάναβη για ιατρική χρήση, ενώ επιτρέπουμε ε, ανενόχλητα άλλα φάρμακα, πολύ πιο Έχει αποδειχθεί η θετική επίδραση της κάναβης ε, ε, νομίζω ότι περισσότερο είναι το ψυχολογικό θέμα της, ε, της ψυχαγωγικής κάναβης και όχι τόσο το, το ιατρικό πρόβλημα. Οι Μεξικανοί έφεραν ε, τη χρήση της μαριχουάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον 20ο αιώνα και μάλιστα ε, τότε είχαν πει στο τέξι ότι όλοι οι Μεξικανοί είναι παλαβοί και είναι το, το χόρτο αυτό που του τρελαίνει. Γι' αυτό και απαγορεύτηκε η παραγωγή. Έχουν περάσει 100 χρόνια και θα πρέπει επιτέλου να έχουμε πιο λογικέ πολιτικέ καλλιέργεια ε, της κάναβης δεν είναι ούτε, ε, ούτε αφύσικο είτε παράλογο. Απλώς υπάγεται στα συμφέροντα μεγάλων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο εξορθολογισμός και η νομοποίηση της χρήσης ε, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής πολλών ασθενών και θα και πραγματοποιήσει ένα βήμα προόδου και συμφιλίωσής μας με τη φύση τους προγόνους μας και τη ζωή. Γιατί η καλλιέργεια κανάβεως αποτελεί τμήμα της παράδοσης όλο χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισπανίας μεταξύ άλλων με κλιματικές ε, αλλαγές, ε, συνθήκες πολύ ευνοϊκές για την καλλιέργεια αυτού του φυτού. Η αηφόρος καλλιέργεια λοιπόν ε, με σεβασμό της φύσης δίνει μια ελπίδα για την υγεία των περιβάλλων, αλλά και πολλές αγροτικές ζώνες του, της Νοτιού Ευρώπης που χρειάζονται κατεπηγόντως ένα παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στην περιβαλλοντική καλλιέργεια και σε μια διαφορετική αντίληψη της ζωής. Χρειαζόμαστε περισσότερη ουσιαστική κυριαρχία και γι' αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο τους πόρους που μας δίνει η ίδια η γη. Ευχαριστώ. Κύριος Πεντιτσίνη. Grazie, grazie Presidente. Eh, anche noi appoggiamo questa σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ε, συνυπογράφουμε αυτήν, ε, την, ε, αυτό το ψήφισμα γιατί πιστεύουμε πως πρέπει να επιτευχθούν κάποιοι στόχοι σε αυτό το τομέα αλλά για να επιτευχθούν πρέπει να αποσαφηνίσουμε δύο πολύ θεμελιώδη πράγματα. Βλέπω πως υπάρχει συζήτηση και στη χώρα μας υπάρχει και επικρατεί μια σύγχυση γιατί γίνεται πολύ χειραγώγηση. πρώτο είναι να διακρίνουμε ανάμεσα στην κάναβη και την ε, ε, ε, θεραπευτική κάναβη, δηλαδή καναβινόλη από καναβιδιόλη. Καναβινόλη είναι η ψυχο... ψυχοτρόπα ουσία, ενώ στην καναβιδιο... καναβιδιόλη δεν υπάρχει αυτή. Είναι η θεραπευτική ουσία. Τώρα το να παραγωγή... Ε, υπάρχει θέμα ε, αγροβιομηχανικής παραγωγής γιατί είναι πέραν της συζήτησης οι, οι θετικές επιπτώσεις των ε, καναβινοειδών στην θεραπεία χρόνιων πόνων, στην ε, άμβλεση των συμπτωμάτων της κλήρησης κατά πλάκας και τα λοιπά και τα λοιπά έχουν, έχουμε επιστημονικές αποδείξεις. Ε, ωστόσο, στην Ιταλία, εφόσον ο καθένας δίνει παραδείγματα από τη χώρα του, το Ανώτατο Συμβούλιο Υγείας ε, με βάση τον μύθο του Υπουργείου Υγείας ε, έχει εκφραστεί και συστήνει να ε, προστρέξουμε στην αρχή της προφύλαξης γιατί δεν υπάρχουν αρκετές λέει επιστημονικές μελέτες για, ιατρικά, τις ιατρικές ιδιότητες της κανάβεως. Όμως πρέπει εδώ να τονίσουμε άλλο είναι η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης σε σχέση με τη χρήση των light καναβινοειδών δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον υγιή πληθυσμό και κάτι άλλο είναι το να λέμε την εφαρμογή των, ε, ε, της χρήσης για ασθενείς, δηλαδή με θεραπευτικό σκοπό. Σε αυτήν την ε, περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αρχή της προφύλαξης, να γίνουν καλύτερα είναι οι φάσεις μελέτης, οι φάσεις 1, 2 και 3, δηλαδή να μελετηθεί ποιος είναι ο αντίκτυπος αυτών των νοσιών, αυτής της ουσίας στα ζώα, καταρχάς και αν μετά στους ανθρώπους από την άποψη της τοξικότητας και δεύτερον της αποτελεσματικότητας. Ε, πρέπει δηλαδή να είναι ε, διακριτά αυτά τα δύο πλαίσια και έτσι να είναι πιο σαφές ποια είναι η στάση ε, που πρέπει να κρατήσουμε σε σχέση με το νομοθεσία που θέλουμε εδώ να συστήσουμε και καλούμε την Επιτροπή να κάνει δράση στήριξη στην έρευνα, στην ανάπτυξη, την έγκριση, την εμπορευματοποίηση, την φαρμακοεπαγρύπνηση αλλά και την πρόληψη της κατάχρησης αυτής της ουσίας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα, ε, κυρία Σαϊπέρεκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και στην Ολλανδία γίνεται μια συζήτηση ειδικά εντός του ΣΕΝΤΕΑ, γιατί βεβαίως η πολιτική έχει μείνει πίσω. Τι μιλάμε για χρήση ενός φαρμάκου από ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι και δεν θα περιμένουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή μια χώρα αρχίζουν για να ανακουφίσουν τον πόνο τους. Και αν δεν μπορούν νόμιμα θα το πάρουν παράνομα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το τι είναι το σωστό. Πριν όμως πούμε ότι κάτι είναι καλό, πρέπει να το ερευνήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς είμαι υπέρ της ε, σωστής ε, διαδικασίας. Ε, και βεβαίως το θέμα δεν είναι να πει η Ευρώπη τι είναι καλό και τι όχι, γιατί είναι και θέμα των ασθενών. Συμφωνώ λοιπόν με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γιούζο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Η κάναβης είναι ένα φυτό που προκαλεί παρεστήσεις. Με επιζήμια αποτελέσματα στον άνθρωπο. Και δίνουμε μάχη να μην καταναλώνεται ε, για ψυχαγωγικούς λόγους, αλλά ε, και θα είναι τρομερό να το αφήνουμε ελεύθερο και ο καθένας θα μπορεί να το χρησιμοποιεί. Αλλά απ' την άλλη έχουμε κάποιου ασθενεί με χρόνιου πόνου που έχουν ως μοναδική λύση τη χορήγηση κάναβε, ή ε, παραγόγων κάναβης, αλλά μόνο μετά από συνταγογράφηση. Το πρόβλημα μου είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αρκετή έρευνα για να βελτιωθούν τέτοιου είδου θεραπευτικέ αγωγέ. Το πρόβλημα είναι ότι σε κάποιε ε, χώρες όπως τη δική μου, χρειάζεται ο ασθενής να προσφύγει σε λαθρεμπόρους ναρκωτικών για να βρει το φάρμακο. Εμείς ε, δεν θέλουμε να είναι ελεύθεροι καναβής για όλους, να μπορούν όλοι να την καλλιεργούν στο μπαλκόνι τους, στο σπίτι τους. Αλλά να κάνουμε κάτι θετικό για την υγεία των ε, Ευρωπαίων. Και η κάναβης για ιατρικούς σκοπούς καλό θα είναι να αποτελεί αντικείμενο έρευνας, αυστηρού ελέγχου και πάντα να χορηγείται μετά από συνταγογράφηση ιατρού. Σε αυτό συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Δεν βλέπω κανέναν. Ο κύριος Μιχόκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συζήτηση αυτή για να πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρεται και στο ψήφισμά σας. Η διάκριση μεταξύ της ψυχαγωγικής χρήσης ε, της κανάβεως και της ιατρικής χρήσης της κανάβεως. Η κάναβης καλύπτεται από διεθνείς συμβάσεις που είναι και ο κρογωνιαίος λήθος για την πολιτική της κατανάλωσης κανάβεως και θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Και μάλιστα οι συμβάσεις αυτές οι διεθνείς απαγορεύουν την χρήση ε, κανάβες για ψυχεί, αλλά την επιτρέπουν για ιατρικού σκοπούς. Και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση μεταξύ ψυχαγωγική χρήση και ιατρική χρήση φαρμακευτικής. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρμοδιότητα να επιληφθούμε τις χρήσεις της κάναβης από άποψη ποινική. Απ' την άλλη θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την δημόσια υγεία. Αλλά για θέματα δημόσια υγεία δεν έχουμε αρμοδιότητα. Απλώ στηρίζουμε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράσουν πρώτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Απλώ μπορεί με κάποια μέτρα να στηρίξει τη δράση των κρατών μελών. Και στο παρελθόν είχαμε και διαφορετικά μέσα ε, χρηματοδοτικά για την πρόθεση της έρευνας στον τομέα αυτό. Έχουμε ακόμη κάποια χρηματοδοτικά μέσα που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδου έρευνα. Για τα θέματα της έγκρισης, καλύτερα να σας μιλήσει ο συνάδελφος από τη Γενική Διάθεση Υγείας. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνατε. Σίγουρα η φαρμακευτική κάναβη ή η κάναβη για ιατρικούς σκοπούς δεν είναι σαφώς προσδιορισμένη έννοια και έχετε διαφορετικές ερμηνείε. Όταν όμως μιλούμε για φάρμακα που είναι παράγωγα καναβινοειδών, τότε μιλούμε για ε, προϊόντα που εγκρίνονται για ιατρική χρήση. Και από αυτή την άποψη έχουμε νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καταρχήν ε, είναι αρκετά ανοιχτό για να περιλάβει και φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν ως δραστική ουσία ένα καναβινοειδές. Οπότε θα εμπέσουν τέτοια προϊόντα στο ε, σύστημα έγκρισης, είτε το εθνικό είτε το κεντρικό. Όπως ανέφεραν κάποιοι ευρωβουλευτές, έχουμε ένα προϊόν αυτή τη στιγμή που έχει λάβει άδεια κυκλοφορία σε πολλά κράτη-μέλη με την διαδικασία της αμοιβαίας αναγνώρισης. Κάτι που δείχνει ότι η διαδικασία έγκρισης ή αδειοδότησης μπορεί να καλύψει τέτοιου είδους προϊόντα, παράγωγα της κάναβης. Έχουμε πολλές σπάνιες νόσους και σε τέτοια είδους θεραπευτική αγωγή αναφέρονται και τα καναβινοειδή ε, πιθανά φάρμακα για χρήση, αλλά δεν έχουν εγκριθεί ακόμη για σπάνιες νόσους. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στις άδειες ε, την υποχρέωση ποιότητας ε, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας και να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις παρενέργειες τέτοιων φαρμάκων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επαρκή έρευνα για να ζητήσουμε μετά από εταιρείε να παρασκευάσουν τέτοια προϊόντα. Θέλουμε επαρκείς αποδείξεις, γιατί το σύστημα έγκρισης που εφαρμόζουμε στηρίζεται σε τεκμήρια, σε αποδείξεις και χρειαζόμαστε και αυστηρή παρακολούθηση και έλεγχο σε ό,τι αφορά τέτοια προϊόντα. Έχουμε λοιπόν τις διατάξεις ε, και το νομοθετικό πλαίσιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων οργανισμών. Έχουμε τον οργανισμό, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τροφίμων ή τον οργανισμό ΤΡΑΚ για την ανταλλαγή πληροφοριών για τη χρήση φαρμάκων. Και εκεί θα πρέπει να δούμε τα τις προδιαγραφές ποιότητας σε σχέση με τη συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι ενδιαφέρουσα η κάναβης, αλλά για να, δοθούν, για να δοθεί έγκριση η άδεια για τέτοια προϊόντα θα πρέπει να στηριζόμαστε σε αδειάστα επιστημονικά κριτήρια και να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σμιτ. Οπότε τελείωσε εδώ πέρα η συζήτηση για το θέμα αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι 4 Ιουλίου στις 11 η ώρα είναι η προθεσμία για τροπολογίες και μάλλον θα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος τον Οκτώβριο στην Επιτροπή μας. Περνάμε τώρα στην ε, προστασία καταγγελόντων παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Ναι, ναι. Εξετάζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης και Δίνω τον λόγο πρώτα στον εισηγητή μας, τον κύριο Μαρσή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος συμμετέχουν σήμερα πέρ του γενικού συμφέροντος. Ε, χάρη σε αυτούς πολλά σκάνδαλα σε σχέση με παράνομες πρακτικές έχουν αποκαλυφθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο πολύ συχνά ακόμα και σήμερα διώκονται, κρίνονται, ε, καταδικάζονται ε, και στις ευρωπαϊκές χώρες τις δικές μας. Α ε, ας θυμηθούμε τον Αντουάν Ντελτούρ για τα Λουξ Λίξη, την Αν Μαρή Καστερέ για την υπόθεση του ε, μολυσμένου αίματος, τη Σεσίλ Μπουσιέ για την ε, κακομεταχείριση αναπήρων παιδιών. Δεν μπορούμε παρά να δούμε, διαπιστώσουμε ότι δεκάδες δημοσιογράφοι απειλούνται επίσης και μάλιστα ορισμένοι καταδικάζονται και ακόμα και ορισμένοι βρίσκονται πίσω από τα, τις φυλακή στα σίδερα επειδή ε, έκαναν την ερευνητική τους ε, δουλειά και τελικά προσπάθησαν να προστατεύσουν το κοινό συμφέρον στο πλευρό των ε, μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Η προστασία λοιπόν αυτών των ανθρώπων είναι ακόμα πιο σημαντική γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί συνήθως διαπράττουν μια επαγγελματική αυτοκτονία εφόσον μια μέρα έχουν το, θα, βρουν το θάρρος για να αποκαλύψουν τι συμβαίνει. Είναι λοιπόν ε, ουσιώδες το να καλύψουμε αυτό το κενό το νομικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σήμερα οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος δεν χαίρουν καμίας πραγματικής προστασίας μέσα στο κοινοτικό δίκαιο και ακόμα χειρότερα η πρόσφατη οδηγία για το απόρριτο των ε, ε, ε, το επιχειρηματικό έρχεται να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την ε, κατάστασή τους καθώς και τους δημοσιο... των δημοσιογράφων καθώς τους καθιστά πιο ευάλωτους δικαστικά. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο ανησυχούμε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα γιατί ε, συχνά και το γνωρίζετε αυτό στους τομείς της υγείας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων ή της προστασίας των ζώων ξεσπούν σκάνδαλα. Και γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που μπορώ να συντάξω γνωμοδότηση επί του θέματος αυτού στο όνομα της Επιτροπής μας ε, του Περιβάλλοντος. Τι συμβαίνει λοιπόν η πρόταση της οδηγίας της Επιτροπής ε, φυσικά αποτελεί ένα βήμα μπροστά ε, και χαίρομαι γι' αυτό. Ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, διότι προβλέπει ένα πλαίσιο προστασίας των πιο ευάλωτων ανθρώπων, δηλαδή που βρίσκονται σε μία σχέση εργασιακή και άρα σε σχέση σε σχέση ε, ανώτερου ή κατώτερου υφισταμένου υπαλλήλου. Άρα λοιπόν θα μπορεί να δεχτεί πιέσεις από τις δημόσιες αρχές τις οποίες εργάζεται, αλλά θα πρέπει εκεί να προστατεύεται και θέλουμε να υπάρχει και μια εθνική αρχή σήμανσης που είναι σημαντική για να μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, σε αυτή μας ε, την προσπάθεια. Όμως την γνωμοδότησή μου προτείνω να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Ε, θέλω να προσθέσουμε αυτά τα δύο επίπεδα, δηλαδή ένα επίπεδο σήμανσης και προστασίας ευρωπαϊκή Πιστεύω όντω πω πολλέ υποθέσεις μας ε, δίδαξαν ότι τα κράτη δεν είναι πάντοτε στην καλύτερη θέση για να ασχοληθούν με τα πιο λεπτά ζητήματα. Γι' αυτό, για να εγγυηθούμε μια πραγματική προστασία στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και να ενθαρρύνουμε ε, τις αποκαλύψεις τους, προτείνω στη γνωμοδότησή μου τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προστασίας των Μαρτύρων Δημοσίου Συμφέροντος. Ε, αυτή η υπηρεσία θα παρέχει ε, απευθείας πρόσβαση στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, ενημέρωση, ανατολισμό των ε, δυνητικών μαρτύρων ώστε να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αλλά θα αποτελεί και ένα πραγματικό ε, διάβλο ε, ενημέρωσης αλλά και προστασίας απόλυτης αυτών των ανθρώπων ενάντια σε αντίπεινα. Αυτή η υπηρεσία θα μπορεί να έρθει σε επαφή με τις εθνικές αρχές, όπως ε, περίπου και η υπηρεσία καταπολέμησης των απατών ή οι ευρωπαϊκές ε, αρμόδιες αρχές θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα εθνικά κράτη, ώστε να λάβουν τα μέτρα και τις απαραίτητες, να προβούν σε απαραίτητες κυρώσεις. Σκέφτομαι, ας πούμε, επίσης την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Όλαφ ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση που περιλαμβάνεται σε αυτήν ε, την ε, γνωμοδότηση. Επιπλέον θέλησα να διορθώσω κάποιες ε, νομικές αδυναμίες και κενά που υπάρχουν σε αυτήν την οδηγία και μπορεί να αποδυναμώσουν την προστασία των μαρτύρων. Θέλω λοιπόν να δούμε, να προστατευτούν οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν όχι μόνο παρανομίες αλλά και αντίθετες προς το κοινό συμφέρον ή στους στόχους του δικαίου, γιατί συχνά το όριο της νομιμότητας είναι λεπτό και στα περισσότερα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν προσφάτως οι υπεύθυνοι βρίσκονται σε μια φαιά ζώνη από άποψη δικαίου. Προτείνω επίσης, και αυτή είναι η τρίτη μου πρόταση κλειδί, να διευρυνθεί το πεδίο προστασίας στο σύνολο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και να εκπεκταθεί η προστασία στους υπαλλήλους των ευρωπαϊκών εταιριών που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας ή ακόμα και στους υπαλλήλους ε, και συνεργαζόμενος των ευρωπαϊκών θεσμικών ιδρυμάτων ή των ευρωπαϊκών οργανισμών χωρίς τους οποίους πολλά σκάνδαλα δεν θα είχαν μπορέσει να αποκαλυφθούν. Δεν χρειάζεται να σας τα παραθέσω όλα, αλλά πρόσφατα είχαμε το προβλήματα για την ηλεκτρική αλληλεία, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, για τη γλυφοσάτη και ένα σωρό θέματα όπου οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν μιας προστασίας. Και επίση στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχει και ένα, μια πρόταση που περιορίζει ίσως το, την προστασία. Δηλαδή δημιουργία μία ιεραρχίας που υποχρεώνει τους μάρτυρες να απευθούν στην εσωτερική, στον εσωτερικό διάβλο ενημέρωσης μέσα στο πλαίσιο της εταιρεία. Εάν υποχρεωθεί να το κάνει αυτός αυτό ο μάρτυρας, αποθαρρύνουμε ε, τον, την αποκάλυψη σκανδάλων, αλλά ε, ε, μπορεί επίσης να επιδεινώσουμε την κατάστασή του, την πρακτική, γιατί μπορεί έτσι να εκτεθεί σε κίνδυνο ε, κυρώσεων ή επαγγελματικών αντιπίνων. Οπότε προτείνω απλά να καταργήσουμε αυτή του είδους την ιεράρχηση και να επιτρέψουμε στον μάρτυρα ε, δημοσίου συμβέροντος να απευθυνθεί χωρίς όρους και ανάλογα με τη δική του επιλογή στους εσωτερικού διάβλους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς και έτσι να τους εγγυηθούμε μια, ένα πραγματικό δικαίωμα αποκάλυψης προς ε, δημοσιογράφους ή ΜΚΟ που ειδικεύονται στην προστασία των μαρτύρων. Ε, τέλος, έχω προτείνει διάφορα, πολλές τροπολογίες για τη βελτίωση συγκεκριμένα της εμπιστευτικότητας και τα, ε, των δικαιωμάτων των μαρτύρων δημοσίου σε όλα τα επίπεδα ώστε να ε, προτείνουμε μέτρα ε, συλλογικά που μπορούν να λάβουν οι αρχές, αλλά και για την προστασία των ενδιάμεσων ανθρώπων που μπορεί να αναμειγνύονται στην αποκάλυψη των πληροφοριών. Αυτή η οδηγία είναι μια οδηγία που ακολουθεί ε, την οδηγία για το τον το χαρακτήρα των επιχειρήσεων Και θα ήθελα λοιπόν να μπορέσουμε να έχουμε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής μας ε, που να είναι πραγματικά χρήσιμη. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτος ο κύριος Τουρκάνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας πω ότι χαίρομαι για το ότι η νομοθετική διαδικασία λειτουργεί ικανοποιητικά. Γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι για το ότι είχαμε δύο ψηφίσματα πέρσι για την προστασία των καταγγελόντων και τον ρόλο τους στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ήμουν σκιώδη εισηγητής για την πρώτη από αυτές ε, και χαίρομαι που είμαι και ε, και για το δεύτερο τέτοιο έγγραφο. Είναι ένα λογικό και ισορροπημένο κείμενο. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο για να μπορούμε να προστατεύουμε τους ε, καταγγέλλοντες. Νομίζω ότι κανείς ε, δεν έχει ξεχάσει τα Panama Papers, το Wikileaks, όπου βλέπουμε ακριβώς ποια σημασία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ο νόμος να τηρείται σωστά. Και μιλάω εδώ πέρα για τα ύδατα, το έδαφος, ζωοτροφές, τρόφιμα λοιπά. Πράγματα που αφορούν την Επιτροπή μας. Παρακολουθήσατε να, τη δουλειά του κύριου Ομαρζή. Να σας πω κάποια πράγματα που επεσήμανα. να αναφερθώ στην σχετική υπηρεσία. Θεωρώ εδώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αναφτιάξουν τις δικές τους ε, αρχές. Από την άλλη, αυτό θα σήμαινε επιπλέον κόστος ε, και ε, γραφειοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να μειώσουμε. Αφετέρου όμως θα ενθαρρυνθεί περισσότερο κάποιος ε, καταγγέλων να καταγγείλει σκάνδαλα κάπου πιο κοντά αντί να απευθυνθεί σε ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είναι ε, δύσκολο να εμπλακούν ε, τρίτοι εδώ. Τρίτοι οι οποίοι δεν έχουν άμεση γνώση του εν λόγω σκανδάλου. Η Κομισιόν δεν μπορεί να επιβάλλει τιμωρίες. Ε, θεωρώ όμως ότι κάθε κράτος μέλος έχει ε, κάποιες ε, σχετικές διατάξεις στην νομοθεσία του. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Τσέλντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτζή για τη δουλειά που έχει κάνει. Ως Ιρλανδοί Ξέρω ότι στην χώρα μου ε, χρησιμοποιούνται συχνά αντίπεινα κατά των καταγγελόντων για να κρυφτούν διάφορα σκάνδαλα και κάποια θέματα που είναι γνωστά αφορούν και την Επιτροπή μας. Πριν από το πρόσφατο σκάνδαλο με το κρέας αλόγου που αποκάλυψαν πρώτα οι επιθεωρητές τροφίμων το 2013 είχε συλληφθεί μία Ιρλανδή δημοσιογράφος επειδή δεν αποκάλυπτε τις πηγές της για τις ατασταλίες στην επεξεργασία βοηου κρέατος. Ε, πρόσφατα άλλαξε η νομοθεσία, αλλά μόνο μία μειοψία κρατών μελών έχουν νομοθετήσει προστασία των καταγγελόντων, κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει ότι έχουμε κατακερματισμένη προστασία και ανεπαρκή Μπορούμε να έχουμε λοιπόν ε, πολύ διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια τροφίμων ανάλογα με το τι αντιμετωπίζουν οι καταγγέλλοντες όταν αποκαλύπτουν κάτι. Χωρίς να αναφέρουμε βεβαίω την διασυνοριακή φύση πολλών δραστηριοτήτων όταν ακριβώς μιλάμε για αποκαλύψεις που αφορούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πολλά από αυτά θα είχαν αποκαλυφθεί νωρίτερα αν υπήρχε το κατάλληλο νομικό πλαίσιο προστασίας. αυτού βλέπαμε παροδίες της δικαιοσύνης όπως η δίκη LuxLeaks όπου κατέληξαν να δικάζονται οι καταγγέλλοντες για παραβίαση απορρίτου. Ήταν βαρύ το τίμημα λοιπόν, ενώ ο κύριος ε, Γιούνκερ ε, κατέληξε πρόεδρος της ε, Κομισιόν και η PricewaterhouseCoopers πήρε συμβάσεις εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ε, κατέληξα να υπερψηφίσω την οδηγία περί εμπορικού απορρίτου για περιπτώσεις ε, στις οποίες δεν ήταν παράνομο το να αποκρύπτει κανείς ε, Χαίρομαι λοιπόν με την πρόταση της Κομισιόν. Καλωσορίζω την πρόταση του κυρίου Όμαρτζή για την σύσταση μιας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σημείο επαφής για όσους βλέπουν ατασταλίες και θέλουν να τις καταγγείλουν. Επίσης ανησυχώ με την αυστηρότητα των προτάσεων για τους διάβλους καταγγελίας που τελικά ίσως στην πράξη δεν επαρκούν για να προστατεύσουν όσους θεωρούν ότι η εσωτερική καταγγελία στο εσωτερικό ενός οργανισμού δεν επαρκεί. Θα πρέπει λοιπόν το πεδίο εφαρμογή οδηγίας να γίνει όσο το δυνατόν ευρύτερο. Να καλύπτει ολόκληρο το πεδίο της ευρωπαϊκής πολιτικής και δικαίου όταν υπάρχει σοβαρός φόβος για το δημόσιο συμφέρον. Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή για το ότι το βάρος της αποδείξεως όταν κάποιος ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει δημόσιο συμφέρον να πέφτει σε αυτούς οι οποίοι το αμφισβητούν. Και ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητέ ε, που έφεραν αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν βλέπω Άλλο και ο στην αίθουσα. Θέλει άλλος κανεί το λόγο, παρακαλώ. Ουδή. Οπότε η κυρία Μερκάντε Πικέρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους προλαλήσαντες για την ανταλλαγή απόψεων και Ευχαριστώ που παρουσιάσατε τόσο σφαιρικά την ε, οδηγία. Δεν πρόκειται να σας ε, αναλύσω διεξοδικά τα στοιχεία της οδηγίας. Ήταν πολύ εμπεριστατωμένη η εισαγωγή του εισηγητού. Απλώς θα σταθώ στους βασικούς στόχους της οδηγίας μας. Ε, είχαμε πολλά σκάνδαλα πρόσφατα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ιδιαίτερο το ρόλο των καταγγελόντων κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Είδαμε την περίπτωση των LuxLeaks και των Panama Papers. Οπότε σίγουρα οι ε, δεν δραματίζουν ε, κύριο ρόλο στην αποκάλυψη ατασταλιών και παρανομιών. Οι Εθνικέ αρχέ από του δεν μπορούσαν να τι είχαν εντοπίσει χωρίς καταγγελίες τέτοιες παρατυπίες. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει την πρόταση προκειμένου να ε, προστατεύσουμε αυτού του ήρωε που αθέλητα έγιναν ήρωες καταγγέλλοντας και δημοσιεύοντας τέτοιες ε, παράνομες δραστηριότητες και έχοντας το κουράγιο να τις καταγγείλουν. Είναι πολύ έγκυρη πρόταση γιατί αφενός ε, το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας καλύπτει τους τομείς του ενωσιακού δικαίου όπου μία παρανομία μπορεί να παραβλάψει σοβαρά το δημόσιο συμφέρον. Και εκεί ε, η έννοια του καταγγέλλοντος έχει προσθεθέμενη αξία. Και γι' αυτό επιλέξαμε 13 τομείς ε, που περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική προστασία, ασφάλεια τροφίμων, καλή μεταχείριση ζώων, ασφάλεια ζώων και ούτω καθεξής. Και εκεί υποβάλαμε μια σειρά μέτρων για την προστασία των καταγγελών των ε, παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Και όπως είπε ο εισηγητής, ε, υπάρχει ένα ευρύ προσωπικό πεδίο εφαρμογή και υποχρέωση θέσπισης εξωτερικών και εσωτερικών διάβλων για τις καταγγελίες. Και μάλιστα ε, και οι εθνικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν σωστά και να παρακολουθούν, να δίνουν μια συνέχεια στις συγκεκριμένες καταγγελίες. Υπάρχει η σαφής ε, διάταξη βάρος των αντιπίνων και μάλιστα αν τελικά υιοθετηθούν αντίπινα κατά του καταγγέλλοντος ε, προβλέπεται η προστασία του. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του εισηγητού και κάποιων ευρωβουλευτών, εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι εθνικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Γι' αυτό η υποχρέωση θέσπιση εξωτερικών διάβλων θα πρέπει να απευθύνεται στις εθνικές αρχές. Δεν έχουμε επιβάλει εμείς ε, ή θεσπίσει ένα ευρωπαϊκό σώμα, γιατί το να θεσπίσουμε ένα τέτοιο σώμα είναι ουσιαστικά ε, να το επιφορτίζουμε με την ε, διαλεύκανση, την εφαρμογή ή την προστασία των καταγγελόντων και κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήταν παρατραβηγμένο κατά τη γνώμη μας. Ε, ένας ευρωπαϊκός φορέας δεν θα πρέπει να υποκαθίσταται στο ρόλο των εθνικών φορέων και την ανάλυση των μεμονωμένων περιπτώσεων. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι φορείς που ήδη υπάρχουν αναφέρονται, όπως η Όλαφ, που είναι ένας ε, εξωτερικός διάβλος. Επίσης, στον τομέα της ασφάλειας της ναυτιλίας υπάρχει μια ε, τέτοια δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει τέτοιες, ε, τέτοιους εξωτερικούς διάβλους. Οπότε η οδηγία προστατεύει αυτούς που χρησιμοποιούν αυτούς τους εξωτερικούς διάβλους. Δεν κρίναμε όμως σκόπιμο να θεσπίσουμε ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό φορέα για τα θέματα αυτά. Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι ευρωυπάλληλοι καλύπτονται από την ε, ενωσιακή νομοθεσία. Όλοι, ε, όλο το προσωπικό, των, όλοι οι υπάλληλοι των Ηνωμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από τις κατευθυντήρες γραμμές ε, ε, και τον κανονισμό του 2013 και 2014 σε περίπτωση που καταγγέλουν ε, απάτες ε, ή διαφθορά εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε με το νέο εσωτερικό κανονισμό το προστασία για το προσωπικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Με την οδηγία αυτή ενισχύουμε την αξιοπιστία του συστήματος και γι' αυτό θεσπίσαμε και κυρώσει ή πρόστιμα μάλλον περισσότερο, όχι για εκείνους που καταστρατηγούν τα δικαιώματα των καταγγελόντων, αλλά για τους ίδιους τους καταγγέλλοντες που εσκεμένα υποβάλλουν εμ, πληροφορίες και κακόβουλα υποβάλλουν πληροφορίες. Από τη στιγμή βέβαια που καλόπιστα πιστεύουν ότι είναι αληθείς οι πληροφορίες που καταθέτουν προστατεύονται, αλλά όλοι όσοι και εμένα υποβάλλουν κακόβουλες πληροφορίες ε, ε, τιμωρούνται και γι' αυτό αυτή η συμπεριφορά αποθαρρύνεται από την οδηγία. Κύριο Μαρζή, έχετε και πάλι εσείς το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριο Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση που μας έκανε. Και να πω ότι είναι προφανές ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά έχουμε ένα σύστημα με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ως αποστολή να βελτιώνει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιλαμβάνεται και εξετάζει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κρίνει ενδιαφέρουσα μεν, αλλά θεωρεί ότι μπορεί να τη βελτιώσει. Και νομίζω ότι αυτό προβλέπει η εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία των θεσμικών οργάνων μας. Και διαπιστώνουμε ότι πολύ συχνά οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν μια θετική αρχή υπέρ της προστασίας των καταγγελόντων, αλλά έχουν και κάποια κενά. Και από αυτά τα κενά τα παραθυράκια που επιτρέπει η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται παραγωνισμός μερικές φορές των στόχων ή έχουμε και αντίθετα από αποτελέσματα εξαιτία αυτών των κενών που δημιουργούνται, που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Τελικά, διερωτώμε ποιος θέλει περισσότερη Ευρώπη. Εμείς θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Και θέλουμε επίσης μια πιο προστατευτική Ευρώπη. Εξού και η πρόταση. Δηλαδή θέλουμε ένα ευρωπαϊκό γραφείο προστασίας των καταγγελόντων που θα επιτρέπει πραγματικά την προστασία αυτών των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να προστατεύουν τους υπαλλήλου τους. Ε, και δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκτός του πεδίου εφαρμογή αυτού του γραφείου. Γιατί όταν ακούω κάποια καινούργια επιχειρήματα, θυμάμαι τα παλιά επιχειρήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Και τώρα πια έχουμε καταλήξει συμφωνία ότι χρειαζόμαστε και μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Θυμάμαι τα παλιά επιχειρήματα επίσης για την Όλαφ. Τώρα όλοι θεωρούμε ότι η Όλαφ έχει λόγο ύπαρξης και είναι χρήσιμη. Όταν λοιπόν υποβάλλω μια πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Γραφείου Προστασία Καταγγελωμένων προκειμένου να εσαρκώσουμε αυτή την περισσότερη Ευρώπη, δεν θα πρέπει να φοβόμαστε μια τέτοια πρόταση. Κατά του λοιπού, συμφωνώ σχεδόν με όλα τα σχόλια των συναδέλφων. Και όντως, σε καμία περίπτωση δεν παροτρύνουμε ή δεν ενθαρρύνουμε την υποβολή ε, ψευδών πληροφοριών για βάσιμο. Κάτι τέτοιο άλλωστε εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία και ούτε αυτή την ε, κατεύθυνση ακολούθησε εγώ στην πρότασή μου, ενθαρρύνοντα τέτοιε κακόπιστε ε, συμπεριφορέ. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την υποστήριξή του. Είναι περίπλοκη έκθεση, σίγουρα επιδέχεται βελτίωση και καλό θα ήταν η Επιτροπή Περιβάλλοντο να υποβάλει μια ενδιαφέρουσα πρόταση, όσο πιο ενδιαφέρουσα γνωμοδότηση προ την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, γιατί σε τελική ανάλυση και το θέμα του πεδίου εφαρμογή και σχεδόν όλα τα επιμέρους ε, σημεία της οδηγίας αφορούν και αρμοδιότητε τη δική μας επιτροπή. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. 4 Ιουλίου λήγει η διορία για την υποβολή τροπολογιών στις 11 το μεσημέρι και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο. Έτσι, στο ενολομέλη μάλλον του Σεπτεμβρίου. Το τελευταίο θέμα λοιπόν αφορά την εφαρμογή της, της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την οδηγία για τα αζωτούχα. Έχουμε λοιπόν 19 ερωτήσεις. 19. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όπως και να έχει. So in blocks. Uh, Θα τις πάρουμε σε ομάδες, ανάλογα με το θέμα. Καθορισμός ευπαθών ζωνών. Ερώτηση του κυρίου ΕΚ. Τον λόγο έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εσάς και τους βουλευτές για αυτή την ανταλλαγή απόψεων γιατί δεν είναι κάτι καθόλου απλό. Ναι, η ρήπανση των υδάτων ανησυχεί τους πολίτες δικαίως γιατί επηρεάζει το νερό που πίνουν γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε τις σχετικές οδηγίες για τα ύδατα και για τα που αντιμετωπίζουν ακριβώς το ζήτημα της υπερβολικής ε, λίπανσης ε, των υδάτων από τα λιπάσματα και ακριβώς εδώ πέρα θεωρούν και οι επιστήμονες ότι έχουμε αρχίσει να πλησιάζουμε τα ερωτήματα. Ξεκινώντας λοιπόν ε, με τις ερωτήσεις και την ερώτηση του κυρίου Στεφανέκη για το υπάρχουν περιοχές που δεν περιλαμβάνονται πιθανώς ακόμα στις ευπαθείς ε, ζώνες και το τι κάνει η Κομισιόν. Ναι, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι πληροφορίες των κρατών μελών το 2016-2017 φαίνεται να δείχνουν ότι υπάρχουν ακόμα στην Ένωση περιοχές με δυνητική ρήπανση των υδάτων που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες αυτές. Οπότε η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογεί τον καθορισμό την επάρκεια των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα και με βάση αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Κομισιόν ίσως χρειαστεί να λάβει νομική δράση κατά κάποιων κρατών μελών. Μάλιστα, στο παρελθόν κάποια κράτη-μέλη βρέθηκαν στο δικαστήριο όταν διαπιστώσαμε ότι οι καθορισμένες ζώνες δεν περιέλαμβαναν όλη την έκταση που θα έπρεπε. Και αν θέλετε να συνεχίσω, κυρία Πρόεδρε, με άλλες ερωτήσεις. Ναι, ναι, οπωσδήποτε, αλλά να, πω πρώτα τις ερωτήσεις. Η δεύτερη αφορά τον καθορισμό ευπαθών ζωνών, εθνικά σχέδια δράσης ε, της κυρίας Μίλλερ. Αντάξει. Συνεχίστε. Για την ερώτηση της κυρίας Μίλλερ για το αν υπάρχουν κριτήρια στην Κομισιόν για την επαλήθευση των εθνικών σχεδίων δράσης. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με την οδηγία, η Κομισιόν δεν εγκρίνει επισήμως τα σχέδια δράσης των κρατών μελών. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν καθώς έχουν δεσμευτεί να υποβάλουν σχέδια που θα είναι συνεπή με τις διατάξεις και τους στόχους της οδηγίας. Οπότε, πρώτα απ' όλα η οδηγία καθορίζει κάποια στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα σχέδια δράσης. Περιόδους εφαρμογής, ε, κατά τις οποίες απαγορεύεται η λύπανση να διασφαλίζεται η ισορροπημένη λίπανση και βεβαίως συγκεκριμένα ότι γίνεται κοντά στις πηγές του νερού. Κατόπιν η Κομισιόν έχει τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας ε, για να υπάρχει διασφάλιση της εφαρμογής ε, της οδηγίας. Συγκεκριμένα εδώ η Κομισιόν αξιολογεί το εάν οι δράσεις είναι αναλογικές ε, με τα προβλήματα της χώρας, τις επιλογές που έχουν με επιστημονική τεκμηρίωση και αν υπάρχει και δημόσια διαβούλευση και κατόπιν για να διασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή η Κομισιόν ίσως ε, αναλάβει νομική δράση εάν ε, καταλήξει στο ότι τα σχέδια δράσης δεν συμμορφώνονται με τους στόχους της οδηγίας επίσης και η κυρία Λουρίκε Μούλερ έχει και μια σχετική ερώτηση να την απαντήσω και αυτήν. Ναι, αναφέρομαι στην άποψη της Κομισιόν για τον ρόλο των σχεδίων δράσης και αν η Κομισιόν διακρίνει τα μικρά και τα μεγαλα κρατημέλη σε σχέση με την κατάστασή τους. Η απάντηση είναι όχι, δεν κάνουμε διάκριση με βάση την έκταση των κρατών μελών ότι αξιολογούμε τα σχέδια δράσης με βάση τις απαιτήσει, τις οδηγίες και τον στόχο. Ο στόχος είναι η ρήπανση, να προλάβουμε την ρήπανση δηλαδή, στην επικράτεια των κρατών μελών και όπως είπα η οδηγία καθορίζει κάποια ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης. Οπότε πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα σχέδια δράση ε, βεβαίω είναι προσαρμοσμένα στι σχετικέ ε, απαιτήσει ε, που αφορούν και τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει τις ε, ε, συνθήκες που επικρατούν για να λαμβάνουν μέτρα προσαρμοσμένα σε σχέση με άλλες χώρες με πιο ομοιογενεί συνθήκε όμως. Εάν τα κράτη-μέλη το κάνουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, που είναι θέμα που εξαρτάται τελείως από αυτά. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Για αυτά τα τρία πρώτα θέματα θέλει κανείς το λόγο ή να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Χόισλινγκ. Για το πρώτο, η Κομισιόν είπε ότι ε, καταδικάστηκε ένας, ένα κράτος μέλος, ε, είναι η Γερμανία, που είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε νέο, νέα νομοθεσία περί λοιπασμάτων. Τι γίνεται, θα επανεξετάσει εδώ η Κομισιόν για το εάν ε, η νέα νομοθεσία επαρκεί. Τι γίνεται, υπάρχει μια ασάφεια, δηλαδή σας είπανε ότι έχουμε νέα νομοθεσία, είναι όλα εντάξει και δεν υπάρχει καμία επίδραση. Δεν υπάρχει όντως καμία επίδραση γιατί υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες εκθέσεις επικριτικές νομίζω. Δεν ξέρω τι άποψη έχει η Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την δικαστική αυτή απόφαση, χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και μάλιστα το δικαστήριο ακολουθεί τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα κενά στις γερμανικές διατάξεις που εφαρμόζουν κατά την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στην αιτιολογημένη γνώμη. Βέβαια, το δικαστήριο δεν εκτίμηση της αλλαγής στην νομοθεσία του 2017 γιατί σε ό,τι αφορά την ε, διορία που αναφέρεται στην αιτιολογημένη γνώμη εμεί θα, θα βοηθήσουμε τις γερμανικές αρχές ώστε να σεβαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τη δικαστική απόφαση. Μάλιστα, ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα τώρα. Παρακολούθηση της συνητρορύπανσης. Πρόκειται για ερωτήσεις του κυρίου Μπέλετ, της κυρίας Μίλλερ και πάλι και του κυρίου Εκ. Τρεις ερωτήσεις, κύριε Ρώσα. Ε, ε, ερώτηση του κυρίου Μπέλετ για την ανάγκη μεγαλύτερη σύγκληση ό,τι αφορά τη συχνότητα και τον τρόπο παρακολούθησης τη νητρορύπανσης από τα κράτη-μέλη. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που εθετήσαμε το Μάιο, διαπιστώνουμε μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την πυκνότητα του συστήματος παρακολούθησης και τη συχνότητα της παρακολούθησης, κάτι που παρεμποδίζει τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Θεωρούμε σε εκ τούτου ότι υπάρχει δυνατότητα και περιθώριο για περισσότερη ε, σύγκληση της συχνότητας και του τρόπου παρακολούθησης ε, και το επισημαίνουμε στα κράτη-μέλη. Βέβαια, εν μέρει αυτό εξηγείται από τις διαφορές που υπάρχουν στις ε, γεωργικές πρακτικές και τα τοπικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά της γεωργίας. Περνάω τώρα στην ερώτηση της κυρίας Μιούλερ, που ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανισότητες και τις διαφορές όταν συγκρίνουμε τα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεσή μας δεν συγκρίνει την ποιότητα ύδατος ή τις τάσεις ό,τι αφορά την ποιότητα του ύδατος μεταξύ των κρατών μελών. Η συγκρισιμότητα των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών περιορίζεται από τις διαφορές των δικτύων και των στρατηγικών παρακολούθησης της συνετρορύπανσης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, η έκθεσή μας, αλλά και στο έγγραφο εργασία μας, έχουμε απαριθμίσει των αποτελεσμάτων με αλφαβητική σειρά. Δεν έχουμε καμία ιεράρχηση των αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να ενημερώνει για το που βρίσκονται τα κράτη-μέλη ό,τι αφορά την υποχρέωσή του που απορρέουν από την οδηγία και αυτό θα πρέπει να το κάνει με σχετικά ισορροπημένο τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Στέφαν Εκ, σε ποιο βαθμό τέτοια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, συμβάλλουν στην ε, ανάπτυξη αυτόματης δηματοληψίας του ύδατος ε, προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές της οδηγίας για την υδρορύπανση. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης τη παρακολούθηση τη ποιότητα του ύδατο και θα βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση. Η χρήση τέτοιων προγραμμάτων και του ορίζοντα 2020 και του ερευνητικού πλαίσιου υπαριθμών 7 χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν για να στηρίξουν την πρόθεση ε, καινοτόμο λύσεων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του, της ποιότητας του ύδατος και της αυτόματης δειγματοληψίας ή την εφαρμογή της ε, ε, νομοθεσίας για το είδωρ. Στο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο το 7ο εντοπίσαμε κάποια σχέδια και προγράμματα που συμβάλλουν με 76 εκατομμύρια ευρώ για τα θέματα αυτά, ενώ στο ορίζοντα 2020 έχουμε πάντα από 40 προγράμματα με χρηματοδοτική κοινοτική ενίσχυση 65 εκατομμύριων ευρώ και έχουμε 230 εταίρους ε, στα προγράμματα αυτά. Για παράδειγμα, σε ένα σχέδιο έχουμε μια, ένα ε, ε, σύστημα παρακολούθησης σε real time της ποιότητας του ύδατος. Επίσης, σε άλλο πρόγραμμα εφαρμόζει καινοτόμα εργαλεία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδροφόρων οριζόντων και επίσης έχουμε σαν τρίτο πρόγραμμα τη χρήση ρομπότ για την παρακολούθηση της ποιότητας του, ύδατος. Οπότε όντως γίνεται τέτοια παρακολούθηση. Καλώς. Επερώτηση για τα θέματα αυτά. Όχι. Οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα. Αξιολόγηση των γεωργικών πιέσεων ή των πιέσεων από τη γεωργία. Ερωτήσεις του κυρίου Μπέλα, της κυρίας Ράιερ Πύρικ τον κύριο Χαϊτέμα και του κύριο Πρέτο. Ο κύριος Ρώσο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση του κύριου Πέλετ αφορά πώς συμπληρώνουμε και ενισχύουμε την αξιοποίηση ε, των στοιχείων που έχουμε στο πλαίσιο των προτάσεων για τα λοιπάσματα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κανονισμός περί λοιπασμάτων και οι οδηγίες για το άζωτο είναι, ε, ε, είναι παραπληρωματικές ε, η οδηγία για τα λοιπάσματα ορίζει την ε, πρόσβαση στην αγορά για τα λοιπάσματα. Δηλαδή, επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή στους από τα ε, συνηθισμένα λοιπάσματα στα βιολογικά λοιπάσματα και εδώ συμπεριλαμβάνονται υλικά τα οποία εν μέρη ή όχι έχουν υποστεί κατεργασία ώστε να ε, συμπεριλαμβάνουν τα συγκεκριμένα ουσίες. Οπότε η οδηγία για την νητρολίπανση δεν στοχεύει τα οργανικά ε, λιπάσματα, ε, απλά ορίζει περιορισμούς για τη χρήση λιπασμάτων κάθε είδους σε περιοχές που ήδη είναι μόλις, ε, ιδιαίτερα επιβαρημένες από το άζωτο. Ε, συμπληρώνουν λοιπόν η μία την άλλη. Περνάω στις ερωτήσεις της κυρίας Άννης Ράιε Πιέρικ. Καταρχάς ένα σχόλιο για την ε, επιφάνεια, για την ποιότητα της γης και του νερού. Είναι από τις καλύτερες στην Ένωση. Εμείς αναφέρουμε μόνο στοιχεία, δεν αξιολογούμε. Στις κάτω χώρες όσον αφορά το νερό έχουμε 11,8% των σημείων παρακολούθησης πάνω από το κατόφλι των 50 mg ανά λίτρο. Κάτω από το όριο δηλαδή του 2,13 ε, ενώ για τα νερά επιφανείας μόνο 0,6 έχουν ε, συγκέντρωση πάνω από τα 15 mg ανά λίτρο. πρέπει να σημειώσουμε ότι το 60% του, ε, των νερών θεωρούνται ατροφικά, ευτροφικά. Άρα οι κάτω χώρες όπως και άλλα κράτη-μέλη ε, πρέπει ακόμα να προχωρήσουν για να φτάσουν τους στόχους της ε, οδηγίας για το ζωτούχα. Υπάρχει τώρα και μία εντύπωση στην σκατοχώρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για όλα αυτά και ότι θα έπρεπε να έχει κάνει διαφορετική πρόταση για να αντιμετωπίσει τα υπερβολικά μεγάλα, μεγάλες συγκεντρώσεις ζώων. Ε, ε, η οδηγία διαπιστώνει την κατάσταση των υδάτων. Από το 2007 ήδη διαπιστώνεται. Πρόκειται όμως για μέσα επικορικότητας, όπου τα κράτη-μέλη έχουν μεγάλο περιθώριο λιγμού για να αποφασίσουν για τις ε, ε, υγειονομικές τους υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν ήταν υπεύθυνοι η αρμόδια υπηρεσία των κάτω χωρών να ορίσει το σύστημα και να επιβάλλει τη λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Άρα λοιπόν η Κομισιόν ή η Ένωση δεν μπορούν να κατηγορηθούν για τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Μια άλλη ερώτηση ήταν εάν η Κομισιόν ήταν πρόθυμη να σχεδιάσει μια μελλοντική εξαίρεση με εστιασμό στην ιδιαιτερότητα των καλλιεργειών. Ήδη το είδος της ε, ε, καλλιέργειας είναι σημαντική παράμετρος γιατί τα είδη των καλλιεργειών στις εξαιρέσεις θα είναι τέτοια ώστε να απορροφούν παρκές άζωτο. Ας πούμε το, γρασίδι το χόρτο έχει αρκετή απορρόφηση ε, αζότου και άρα λοιπόν ε, μπορεί να ε, εξαιρεθεί. Αν μπορεί να αποδειχθεί ότι άλλες καλλιέργειες σε συνδυασμό με συγκεκριμένες πρακτικές, ε, εδάφη ή κλιματικές συνθήκες επίσης απορροφούν άζωτο και δεν αποτελούν κίνδυνο, φυσικά θα ληφθούν υπόψη. Η χορήγηση της εξαίρεσης σύμφωνα με την οδηγία είναι δυνατή μόνο εφόσον υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αυξημένο κίνδυνο για την ποιότητα των υδάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις ότι η, ε, ε, όλα αυτά γίνονται χωρίς να υπάρχει έκκληση αζότου και φωσφόρου στα, ε, ε, στα ύδατα της περιοχής. Ρωτήσατε για τα, ε, επίσης στην ερώτηση αναφέρονται ποια ήταν τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη. Αυτό που θέλουμε να ε, διευκρινίσουμε ότι αυτό το κριτήριο για το ε, πάυση της χρήσης κοπριάς αφορά, αφορά ε, συγκεκριμένες ε, περιοχές. Έχουμε ξεκινήσει ένα διετές πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει να ορίσουμε ενορμονισμένα κριτηρία ώστε τα λιπάσματα, τα ζωτούχα που εν μέρη ή πλήρως προκύπτουν από κοπριά να χρησιμοποιηθούν σε περιοχές όπου η πληρως προκυπτουν απο κοπρια να χρησιμοποιηθουνται σε περιοχες οπου η ρηπανση των υδάτων δεν ε, υπάρχει και άρα ε, θα υπόκειται στην οδηγία περί αζωτούχων ή άλλων ε, λιπασμάτων. Θα δούμε λοιπόν ποια, υπάρχει, ποια κατάσταση υπάρχει, πόσο έχουν διεισδύσει τα, η, η νητρορύπανση τα ύδατα. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό προκύπτει για, το, για συγκεκριμένο στοιχείο που παράγεται από τη χρήση κοπριάς ε, και πρέπει αυτό να ε, μετρηθεί. Η κατεργασμένη κοπριά εμπίπτει στην ε, υπόλοιπη ε, και εμπίπτει φυσικά στα υπόλοιπα προγράμματα που εφαρμόζονται μέσω της οδηγίας. Γιατί όπως είναι γνωστό υπάρχει ψηλότερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για νητρορύπανση από τα οργανικά αυτά λιπάσματα. Τώρα, άλλη ερώτηση για την πρόταση της Κομισιόν για εξισορρόπηση των, των λιπασμάτων αντί για την εφαρμογή ε, ορίων και κατά πόσο ε, είμαστε πρόθυμοι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσω της αρχής της εξισορρόπησης των λοιπασμάτων που σωστά αναφέρεται, η οδηγία ήδη προβλέπει συγκεκριμένα συστήματα για, την, ε, για τα λοιπάσματα σε συγκεκριμένα αγροκτήματα. Θα πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιούνται στις σωστές όγκους ε, ε, με βάση την επιφάνεια με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βελτίωση ε, της ποιότητας των υδάτων και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η εφαρμογή τους να μπορεί να παρακολουθηθεί και να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές γιατί αυτές έχουν την ευθύνη για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την νομοθεσία. Νομίζω κυρία Πρόεδρε πως κάλυψα όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ε, για την άδεια αίθουσα. Έρχονται και εκλογές. Και συζητάμε εδώ πέρα για τα πράγματα που αφορούν τους ε, γεωργούς και δεν υπάρχουν καθόλου ευρωβουλευτές. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα ε, αν εξηγήσει η Κομισιόν το τι μόλις συζητήθηκε στην Ολλανδία Κάναμε όλα όσα ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη ε, η χώρα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά ε, από όλε τις ε, πλευρές όσον αφορά ακριβώς το καθαρό νερό και τον αέρα και τα εδάφη και έχουμε ακριβώς μεγάλα προβλήματα με εκμεταλλεύσεις που δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν έτσι και ακριβώς ε, υπήρξε και μια μεγάλη συζήτηση στην Ολλανδική Βουλή με τον ε, αρμόδιο Υπουργό και με τους γαλακτοπαραγωγούς για να ε, υπάρξει ένα μεταβατικό μοντέλο στην Ολλανδία, να δούμε το τι είναι δυνατόν και να δούμε επίσης το τι μπορεί να γίνει. Τέλος τα έχω γράψει και στην ερώτησή μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για την Ολλανδία. Γιατί ακριβώς το ζήτησε και το είπε και χτες ο αρμόδιος υπουργό για το τι μπορεί να γίνει στην περίπτωσή μας για να διατηρηθεί ζωντανό και το όραμα αυτό της Ευρώπης και κοιτάω και το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είναι δυνατό να έχουν οι άλλες χώρες νέα νομοθεσία και να έχει μείνει πάλι η Ολλανδία πίσω. Γιατί καμιά φορά λένε οι Γερμανοί ότι έχουν τρελαθεί οι Ολλανδοί. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μας βοηθήσει η Κομισιόν να βρούμε ένα μεταβατικό μοντέλο. Να έχουμε κορυφαίες επιχειρήσεις, ε, κάνουμε τα πράγματα σωστά και ελπίζω πραγματικά να το τηρήσει αυτό η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Uh, director, do you Κύριε Διευθυντά, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Να πω απλώ ότι θέλουμε να βοηθήσουμε και τα κράτη-μέλη αλλά και τις υπόλοιπες χώρες. Και τα, τις και τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Όντως, ε, στις έχουν την υψηλότερη συχνότητα ε, ζωικού κεφαλαίου και επίσης ε, συχνότητα φωσφορούχων και νητρικών αλάτων άνω του μέσου όρου. Ε, αλλά θα συνεργαστούμε και με τι κατοχώρε και με οποιοδήποτε άλλη χώρα μέλος που χρειάζεται βοήθεια. Ευχαριστώ κύριε Πύρεκ. Ευχαριστώ για την απάντηση. Το θέμα ακριβώς όμως είναι η κυκλοφορία την οποία αναφέραμε και το υπόλοιπο ε, σύστημα. Ελπίζω να καταφέρουμε σύντομα να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα και να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκεί. Ευχαριστώ. Έχουμε βεβαίως και... Ο κατεξοχήν κοπρία. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι ακριβώς πρέπει να προσέχουμε λίγο τους ε, αγρότες. Είναι σαφές νομίζω. Να Ακούστηκαν κάποια πράγματα Αυτά. Θα πρέπει λοιπόν οι υποσχέσεις που ε, έχουν γίνει να τηρηθούν. Κυρία Πρόεδρε, δεν μου αρέσουν ε, οι πολιτικές συζητήσεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες, αλλά εδώ πέρα είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και χρόνια πριν από προηγούμενη κυβέρνηση αλλά θέλω τώρα να βρεθεί μια λύση. Να δούμε το τι κάνουν οι Γερμανοί και το τι μπορούμε και εμείς να κάνουμε στον γαλακτοκομικό τομέα. Συμφωνώ μαζί σας πράγματι να τηρηθούν οι υποσχέσεις, αλλά βλέπουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες μας. Εγώ άκουσα την Κομισιόν και θα ήθελε εδώ πέρα να μας στηρίξει ο κύριος Χάιτεμα. Uh, Δεν έχω καταλάβει το Ολλανδικό το, το θέμα. Ε, θέλετε να απαντήσετε πάλι. Όχι. Ας το αφήσουμε λοιπόν προς στιγμή. Κάποιος άλλος για τα θέματα αυτά. Ωραία. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο. ποιότητα νερού. Η κυρία Κάντενμπαχ, Μπόλκεν, Χάιτεμα πάλι και πάλι Στέφαν Εκ. Έχετε τον λόγο, κύριε Διευθύντα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να αφαιρθώ στην ερώτηση της κυρίας Κάντενμπαχ. Μας ρώτησε τι θα κάνει η Κομισιόν για να επιταχύνει την πρόοδο για την χρήση των αζωτούχων και την εισρωή του στα υπόγεια ύδατα γιατί είχαμε μια βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν σε σχέση με την περίοδο 2012-2015. Οπότε, βεβαίω αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, παραδείγματος χάρη μέτρα τα οποία θα αφορούν ακριβώς ε, τι συγκεκριμένες συνθήκες, σχέδια δράσης ε, που θα φτάνουν μέχρι το επίπεδο της αγροτικής εκμετάλλευσης και αποτελεσματικές συμβουλές για να στηρίξουμε τους αγρότες ε, και μηχανισμοί επιβολής ε, και βεβαίως επαρκή σχεδιασμός. Μάλιστα, το 2016 η Κομισιόν ολοκλήρωσε ένα πιλωτικό έργο που ζήτησε το Κοινοβούλιο για να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα αζωτούχα και τα αποτελέσματα που υπήρχαν ε, τα έχουμε στην σελίδα μας ε, και επίσης ε, δίνουμε στήριξη και μέσω του ορίζοντα 2020 για έρευνα και καινοτομία. Επίσης το πρόγραμμα EU Life προωθεί καινοτόμες λύσεις στην ρήπανση όσον αφορά επίσης και την ρήπανση από λιπάσματα στην Γεωργία. Αυτά υπάρχουν στη σελίδα μας. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρχουν τακτικές συζητήσεις στα κράτη-μέλη, στην αρμόδια ομάδα ειδικών και έχουμε και διμερείς επαφές για την εφαρμογή της οδηγίας και ε, οργανώνουμε τακτικά παρουσιάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτομίες. Και τέλος, στην περίοδο που καλύπτει η έκθεση. Έχουμε επίσης κοινή διαδικασία υπαρβάση κατά 100 μελών για να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία. Μία σχετική ερώτηση της κυρίας Κάντενμπαχ αφορά το εάν η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να λάβει υπόψη το ότι δεν θα πρέπει να επιδοτείται η δραστηριότητα που παράγει τόσο ψηλά επίπεδα ζωτούχων γιατί μετά θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε ξανά το νερό για να είναι πόσιμο. Ε, κοιτάξτε, στην ε, πολιτική την ε, αγροτική οι αγρότες που λαμβάνουν στήριξη έχουν τη λεγόμενη πολλαπλή συμμόρφωση. Είναι μια υποχρέωση. Και βεβαίω οι υποχρεώσει αυτέ περιλαμβάνουν και την οδηγία των αζωτούχων. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν γίνονται σεβαστέ οι υποχρεώσει, υπάρχουν ποινέ. Και σε περίπτωση υποτροπή μπορεί να ανασταλεί η χρηματοδότηση τη ΚΑΠ. Έχουμε λοιπόν αυτή την διαχείριση, την πολλαπλή συμμόρφωση για τις υποχρεώσεις ε, που προβλέπει η σχετική οδηγία. Οι σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχουν σύμβουλες σε γεωργούς για ζητήματα που αφορούν την ε, πολλαπλή συμμόρφωση. Επίσης, τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου μπορούν να στηρίξουν σημαντικές επενδύσεις όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης κοπριάς και την ε, μετάβαση στην βιολογική γεωργία. Για τη νέα πρόταση της ΚΑΠ που παρουσιάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες και που είναι επίσης ε, στα χέρια του Κοινοβουλίου για να υπάρχει μια συνέπεια της πολιτικής ε, θα έλεγα η αιρεσιμότητα είναι αυτό το οποίο συνδέει τις πληρωμές με την συμμόρφωση των δικαιούχων με τις περιβαλλοντικές διατάξεις, κλιματική αλλαγή, δημόσια υγεία, ευσοία των ζώων, υγεία φυτών και ζώων. Συγκεκριμένα θα έλεγα ότι υπάρχει και η ενισχυμένη αιρεσιμότητα που πλέον καλύπτει και την οδηγία πλαίσιο για τα αζωτούχα και βεβαίω τις επαρκείς ε, συνθήκες ε, για την ε, βιωσιμότητα των αγροκτημάτων ακριβώς για τα λοιπάσματα. Κατόπιν υπάρχει ένα ερώτημα του κυρίου Τίμο Βόλκεν. Με συγχωρείτε, μου λένε οι διερμηνείς ότι μιλάτε λίγο γρήγορα. Μάλιστα, ζητώ συγγνώμη. Θα μιλήσω πιο σιγά. Οπότε το ερώτημα του κυρίου Φόλκεν αναφέρεται στο ότι ε, πολλές εταιρείες ύδατος αναμειγνύουν τα υπόγεια ύδατα με καθαρά ύδατα για να υπάρχει επαρκής ε, ποιότητα. Το ξέρουμε αυτό σε πολλές περιοχές και κοστίζει. Δεν έχουμε συγκεκριμένες ή συστηματικές ε, πληροφορίες για το κόστος της ανάμιξης ε, υπογείων ε, υδάτων ή πυδάτων από πηγές ε, με καθαρό νερό. Υπάρχουν όμως κάποιες ενδείξεις του υψηλού κόστους που επιφέρει η ρήπανση με αζωτούχο. Παραδείγματος χάρη υπολογίζεται ότι στη Γαλλία οι απώλειες εισοδημάτων λόγω του ευτροφισμού είναι μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων το έτος για τους παράκτιους δήμους και η επιπλέον επεξεργασία του νερού για να γίνει το νερό πόσιμο υπολογίζεται ότι κοστίζει μεταξύ 120 και 360 εκατομμυρίων ευρώ το έτος. Οπότε, η Κομισιόν σκοπεύει να παρακολουθήσει πιο στενά το ζήτημα του κόστους που σχετίζεται με την επεξεργασία του νερού για να μειωθούν τα αζωτούχα, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται στενά με την αρχή «Οριπένων πληρώνει». Είναι προφανές ότι η επίτευξη του στόχου της οδηγίας ε, σχετίζεται στενά με την ...οδηγία ποσίμου ύδατος. Και βεβαίως η οδηγία αυτή ε, όσο πιο καλά εφαρμόζεται τόσο μικρότερο κόστος καθαρισμού θα έχουμε. Επ' αυτή τη σκοπιά η Κομισιόν την 1η Φεβρουαρίου ενέκρινε μια πρόταση για μια αναθεωρημένη οδηγία πόσιμου ύδατος για να βελτιωθεί η ποιότητα του πόσιμου ύδατος και να υπάρχουν ε, οι κατάλληλες οδηγίες και πληροφορίες στους πολίτες. Έτσι θα έχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές. Τα ζωτούχα περιλαμβάνονται ρητός στο παράρτημα 4. Θα πρέπει λοιπόν να είναι διαθέσιμα στους καταναλωτές με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη. Και τώρα έρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Χαΐταμα. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης ευτροφισμού από τα κράτη-μέλη με βάση παραμέτρους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με τα κράτη-μέλη μια διαβούλευση προσπαθώντας να καταλήξουμε σε εναρμονισμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση του ευτροφισμού και στα πλαίσια της οδηγίας για την υτρορύπανση και στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο για το είδωρ. Επιμένουμε ιδιαίτερα στην ανάγκη μεθοδολογιών που θα αξιολογούν ε, σε υδάτινους ε, πόρους ε, τον ευτροφισμό και θέλουμε συγκρίσιμα στοιχεία με παρόμοια είδη συγκεντρώσεων ύδατος. Επίσης υπάρχει η υποχρέωση της προδιαγραφής καλών οικολογικών προτύπων σε ό,τι αφορά ε, φωσφορούχα και νητρικά αλάτα στα κράτη-μέλη. Οπότε τα προγράμματα μετρήσεων ε, με βάση την οδηγία πλαίσιο για το είδωρ να λαμβάνουν υπόψη τις ε, πιέσεις για την ποιότητα του ύδατος. Σε ό,τι αφορά την συναφή ερώτηση του κυρίου Εκ, το κατά πόσο μια κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση του ευτροφισμού χρειάζεται, ήδη απάντησα προς αυτό. Αλλά έχει και ένα δεύτερο τμήμα η ερώτηση. Ποια είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την επαναχρησιμοποίηση του φορτίου φωσφόρου. Η οδηγία για την υδρολιπασία δεν αναφέρεται ε, ρητά στο φόσφορο. Αλλά ε, η αποφυγή της, του ευτροφισμού είναι στόχος και άρα μια καλύτερη διαχείριση της κοπριάς του ζωικού κεφαλαίου θα μετριάσει το φόσφορο και τα νητρικά άλατα Πολλά μέτρα στα εθνικά σχέδια νετρορύπανσης θα βελτιώσουν και τη διαχείριση του φωσφόρου. Γιατί έχουμε πολύ συχνά ειδικά μέτρα για το φωσφόρο όπως ε, προδιαγραφές εφαρμογής φωσφορούχων λιπασμάτων για, το, για τον ε, ορισμό των ευάλωτων ε, ευπαθών περιοχών μητρικών αλάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο φόσφορος που είναι ο βασικός παράγων ευτροφισμού. Αλλά αυτό είναι εμπίπτει στην ε, διαδικασία παρακολούθηση των κρατών μελών και στην οδική πλαίσιο για το είδωρ. Ε, καλύπτουμε και την πίεση του φωσφόρου σε ό,τι αφορά το, την υλοποίηση του στόχου της καλής ε, οικολογικής προδιαγραφής και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα στα πλαίσια το σχεδίο διαχείρισης λεκανών απορροής. Τώρα, αν υπάρχει πρόθεση διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας νητρορύπανης για να καλύπτει και το φόσφορο, προς το παρόν δεν έχουμε τέτοιους σκοπούς. Η οδηγία για την ηθρορύπαση σε συνδυασμό με την οδηγία πλαίσιο για το είδωρ θεσπίζουν ένα επαρκές πλαίσιο ώστε να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τον ευτροφισμό. Πάντως παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τα μέτρα των κρατομέλων στα πλαίσια του ισχύοντο νομικού πλαισίου, ώστε να καλύπτεται και ο φόσφορο στα θέματα του ευτροφισμού και να εφαρμόζονται σωστά τα σχετικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαϊτεμα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Δελγάδο για τις απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχω μια ερώτηση και πάλι για την αξιολόγηση του ευτροφισμού. Πόσο πιστεύετε το κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τα αίτια της ρήπασης. Τα αίτια των φωσφορούχων και νητρικών εκπομπών από τη Γεωργία ή από άλλε πηγές όπως είναι οι μεταφορές ή τα νοικοκυριά ή από τη θάλασσα. Η απο αλλε πηγες οπως οι μεταφορες η τα η απο τη θαλασσα η βορεια θαλασσα για παράδειγμα, μπορεί να είναι πηγή. Και άλλες πηγές εκπομπών φωσφορούχων υπάρχουν ή αζωτούχων που επηρεάζουν την κατάσταση ευθροφισμού. Ε, δεν θέλω να κατηγορούμε τη γεωργία για πράγματα που, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη και να επιβάλλουμε στη γεωργία κάποια μέτρα που τελικά δεν θα έχουν αποτελέσματα γιατί δεν ευθύνεται η γεωργία για όλα. Επίσης, σχέση με προηγούμενη ερώτηση αν γνωρίζαμε καλύτερα τις ροέ θρεπτικών ουσιών σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και γνωρίζοντας καλύτερα τις εκπομπές σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, τότε θα είχαμε καλύτερη ε, γνώση των εκπομπών της γεωργίας και να, θα, δεν θα χρειαζόταν να κατηγορήσουμε άδικα τη γεωργία για πράγματα που δεν ευθύνεται. Υπάρχει πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις και εξολογήσει. Φυσικά υπάρχουν και άλλε πηγέ αζωτούχων. Δεν είναι μόνο η γεωργία παραγό αζωτούχων, αλλά ειδική για την υδρορύπανση μιλάει συγκεκριμένα για τα αζωτούχα που προέρχονται από τη χρήση λιπασμάτων. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή αν τα κράτη-μέλη στα εθνικά προγράμματα για τα θέματα αυτά λαμβάνουν υπόψη και σε ποιο βαθμό τις άλλες πηγές πίεσης ή τις άλλες πηγές ρήπανσης με αζωτούχα. Αναφερθήκατε στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι αποδέκτης και όχι πηγή περισσότερων ζωτούχων. Αλλά όντω υπάρχουν και άλλε πηγέ ρήπανση με ζωτούχα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν είναι μόνο η γεωργία. Πάντω η οδηγία για την ιτρορύπαση όταν εφαρμοστεί σωστά, δεν επιβαρύνει τη γεωργία. Επικεντρώνεται απλώ στην ιτρορύπαση που προέρχεται από τη γεωργία. Οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια καλύτερης ε, συγκέντρωσης στοιχείων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης για τη συγκεκριμένη κατάσταση των ε, συνθήκων, ε, το, της κατάστασης του εδάφους και μάλιστα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης θα μας επιτρέψει να δημορφώσουμε μια καλύτερη εντύπωση για τις εκπομπές που προέρχονται από τη γεωργία σε σχέση με τις άλλες πηγές ρήπανσης. Πύρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να αναφέρω και εγώ στην ερώτηση του κύριου Άιτεμα. Αυτό σχετίζεται στην Ολλανδία με το καθεστώς των αζωτούχων που έχουμε. Αν δείτε, στη δυτική χώρα υπάρχουν πολλά αζωτούχα στο χώμα, αλλά αυτό δεν έχει τόσο πολύ σχέση με την ε, κτηνοτροφία, αλλά περισσότερο με τα ύδατα και την θάλασσα. Και έχουμε διαφορετικά νούμερα. από τις διάφορες αρχές και το ερώτημά μου είναι ακριβώς τι κάνουμε εδώ πέρα, ε, τι κάνει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κινητοποιείται, ε, παρακινείται την Ολλανδία να δώσει τα σωστά νούμερα, δηλαδή που τι οφείλεται στην γεωργία, τι οφείλεται στην βιομηχανή γιατί αυτό είναι αποφασιστικό, γιατί τελικά κάποιοι θα πρέπει να υπομισθούν αυτό το βάρος που είναι μεγάλο. Παρακαλώ. Κοιτάξτε. Γενικώ ε, στηριζόμαστε στα στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Αυτά μας δίνουν στοιχεία για τα φωσφορούχα και αζωτούχα τα κράτη-μέλη και με βάση τα στοιχεία τους ε, και τη συμπίληση των στοιχείων αυτών ε, προβαίνουμε στις δικές μας αξιολογήσεις. Μάλιστα, άλλος κανείς. Οπότε να περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις που αφορούν διάφορα θέματα. Οπότε, κύριε Ρώσα, απαντήστε ξεχωριστά και μετά από κάθε θέμα, αν υπάρχουν συμπληρωματικές ερωτήσεις, να τις ακούσουμε. Κύριε Ρώσα. Ευχαριστώ πρώτη ερώτηση του κύριου Μπέλετ για το ποια είναι τα αίτια της καθυστέρησης της ε, εκτελεστικής εφαρμοστικής έκθεσης. Η έκθεση ε, συνδυάζει πολλά στοιχεία περιποιότητας ε, από 28 κράτη και κανονικά αναμενόταν από τον Ιούνιο του 2016. Μόνο 12 χώρες όμως μέχρι τότε είχαν σεβαστεί την προθεσμία και μάλιστα για τέσσερις από αυτές δεν είχαν δοθεί αρκετά στοιχεία που αναβλήθηκαν και αργότερα. 19 χώρες δεν έδωσαν στοιχεία ε, καθόλου ή έδωσαν ακατάλληλα στοιχεία. Τα περισσότερα από αυτά συμπλήρωσαν τις πληροφορίες το 2017, οπότε το σύνολο των πληροφοριών για την έκθεση έφτασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καθυστερημένα, τον Οκτώβριο του 2017. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιες καθυστερήσεις στην επόμενη περίοδο υποβολής αναφορών κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2020. Να περάσω στην επόμενη ερώτηση. Καλώς. Περνάμε στην ερώτηση του κυρίου Βόλκαν που ρωτά τους περιορισμούς της οδηγίας για, την ητρορρύπα σε σχέση με το γεωργικό μοντέλο που χρειάζεται για παραγωγή χαμηλών θρεπτικών ουσιών. Και ποια είναι τα μέτρα εκτός της οδηγίας που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της οδηγίας. Η οδηγία για την νητρορύπαση ενθαρρύνει ε, την χρήση βιώσιμων γεωργικών μοντέλων με βάση την ισορροπία των θρεπτικών ουσιών και απευθύνει έκκληση για μείωση της νητρορύπανσης, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιφερειών και των χωρών μελών. Ένα βασικό στοιχείο της οδηγίας είναι ε, η αρχή της ισορροπημένης λίπανσης. Με βάση αυτή την αρχή, οι θρεπτικές ουσίες που, επιβάλλονται που ε, εφαρμόζονται θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανάγκες των καλλιεργιών και αυτό ισχύει και για τα οργανικά και για τα ανόργανα λιπάσματα. Οπότε η οδηγία μας βοηθά να υλοποιήσουμε ή να οδεύσουμε στην πορεία της ε, βιωσιμότητας. Βέβαια, τα μέτρα της οδηγίας αυτής θα πρέπει να συμπληρωθούν από τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν τα μέτρα τους στα πλαίσια άλλων πολιτικών, όπως της πολιτικής για την οδηγία, για την ποιότητα του ύδατος ή τη, στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής. Μόνο με μια συνεκτική προσέγγιση συμπληρωματική θα αποφύγουμε ε, επιζήμιο αποτέλεσμα για τη βιασιμότητα και θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τις επιδοτήσεις και υπέρ της βιωσιμότητας. Οπότε θα πρέπει να στραφούμε προς γεωργικά μοντέλα που χρησιμοποιούν λιγότερες εισρωές, για παράδειγμα βιολογική γεωργία, ή άλλα γεωργικά μοντέλα που χρησιμοποιούν περισσότερο φυσικά και όχι τεχνητές, φυσικές και όχι τεχνητές εισρωές και περιορίζοντας φυσικά και την ητρορύπανση ταυτόχρονα. Διαφέρετε κανείς, όχι, συνεχίστε. Α, μια στιγμή, κύριε Διευθυντά, η κυρία Τελαή. Ευχαριστώ. Δεν πίστευα ότι θα έπρεπε να παρέμβω, αλλά τα όσα άκουσα με κάνουν να ε, παρεμβαίνω. Νομίζω ότι πρέπει να πάψουμε να αντιπαραθέτουμε τα διάφορα αγροτικά μοντέλα μεταξύ τους. Σε λίγο θα ασχοληθούμε με τη δραστική ουσία του χαλκού που χρησιμοποιείται στη βιολογική παραγωγική. Έχει λιγότερο αντίκτυπο ε, για το περιβάλλον και την υγεία από ότι ένα προϊόν συνθετικό. Ε, πρέπει λοιπόν να πάψουμε να τσακωνόμαστε για τις μεθόδους και για τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε τα συνθετικά προϊόντα τα, δεν είναι τόσο βία και τόσο βλαβερά όσο η φύση, ε, όσο αυτό που έχει πολλές φορές παράγει η ίδια η φύση. Οπότε ας μην... Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχολεία σας. Α, να απαντήσω. Γιατί χαίρομαι με το σχόλιο αυτό. Γιατί δεν έχω στόχο ε, να θέσουμε τη μία μορφή γεωργίας ε, ενάντια στην άλλη. Λέμε ότι εκεί όπου υπάρχουν περιοχές που έχουν ήδη ρήπανση από πάρα πολλές ε, εισφορές ε, στοιχείων ε, στο έδαφος είναι ακριβώς να δούμε τις πηγές εκείνες και τους τρόπους παραγωγής που ακριβώς θα μειώσουν αυτές τις πηγές ρήπων. Βεβαίως όλες οι μορφές γεωργίας μπορούν να προσφέρουν στην βιωσιμότητα. Κάποιος άλλο μάλιστα. Συνεχίστε, κύριε Διευθυντά, με την ερώτηση κυρίας Μίλλερ. Κυρία Μίλλερ, για το ποιε διαδικασίες επί παραβάση είναι ακόμα ανοιχτέ και αν θα υπάρξουν νέε δράσει κατά κρατών μελών για την οδηγία των αζωτούχων. Απλά, αυτήν τη στιγμή υπάρχουν έξι διαδικασίες επί παραβάση για τα ζωτούχα σε εξής χώρες. Μία στο Βέλγιο για τη Βαλονία, στη Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία και Σλοβακία. Δύο επίσης ανοιχτές έρευνες που αφορούν την Ισπανία και τον Ομόνο Βασίλειο. Και όπως είπα η Κομισιόν αυτή τη στιγμή αξιολογεί περαιτέρω την τρέχουσα εφαρμογή της οδηγίας με βάση τα τελευταία δεδομένα και ίσως αναλάβει περαιτέρω νομικές ενέργειες εάν απαιτηθεί. Εάν όχι, περνάμε στη δεύτερη ερώτηση της κυρίας Μίλλερ. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο σχετικές ερωτήσεις, μία της κυρίας Μίλλερ και μία του κυρίου Εκ. Ε, να τις απαντήσω μαζί. Η δεύτερη ερώτηση της κυρίας Μίλλερ είναι για τα στρατηγικά σχέδια της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, θα είναι ευκαιρία για περιφερειακή εφαρμογή και μια απλοποίηση ενώ η ερώτηση του κυρίου ΕΚ είναι το εάν η εφαρμογή της οδηγίας περί αζωτούχων ελήφθη υπόψη στην προετοιμασία της κοινή γεωργικής πολιτικής και αν η σωστή εφαρμογή θα είναι ένας από τους όρους εξάντε στο στρατηγικό σχέδιο και θα απαντήσω μαζί. Το στρατηγικό σχέδιο βεβαίως θα πρέπει να λάβει υπόψη τα υποχρεωτικά μέτρα του σχεδίου δράσης που επιβάλλονται στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και θα πρέπει να συμπληρωθεί με επιπρόσθετα εθελοντικά μέτρα έχοντας πάντα κατά νου την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Όπως είπα και πριν, η εφαρμογή της οδηγίας αυτής περιλαμβάνεται στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης και έχουμε αναγγείλει ενισχυμένη αιρεσιμότητα μετά το 2020 που θα περιλαμβάνει διατάξεις που θα συνδέουν άμεσα την, τον σεβασμό των απαιτήσεων αυτών και των άμεσων πληρωμών στους γεωργούς και των ορθών αγροπεριβαλλοντικών πρακτικών. Όπω είπα, αυτές οι διατάξεις έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την ύπανση από ζωτούχα και να, μειώσουν, να βελτιώσουν την εφαρμογή τη οδηγία. που υπάρχουν τώρα στην ενισχυμένη αρισιμότητα. Το ένα είναι το εργαλείο βιωσιμότητα για τα λοιπάσματα και μια νέα διάταξη που απαγορεύει την λίπανση της πιο ευαίσθητε περιόδου. και έτσι τα νέα στρατηγικά σχέδια θα πρέπει να εγκριθούν από την Κομισιόν. Πρόκειται για μια πρόοδο σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο όπου α, τα κράτη-μέλη απλά κοινοποιούσαν τι επιλογέ του στην Κομισιόν. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ για την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την συνέπεια μεταξύ των επιλογών και των αναγκών που προκύπτουν από την αδαγία περί ή, συγκεκριμένα, γενικότερα από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Θα κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για το θέμα αυτό, το οποίο είναι το εξής. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου τους επόμενους ε, μήνες ε, θα πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε την πλήρη συνέπεια στην άσκηση της, ε, πολιτικής, ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών πολιτικών όσον αφορά ακριβώς την στήριξη των γεωργών για να περάσουμε σε ένα πραγματικά βιώσιμο ε, γεωργικό τομέα. Ξέρω πως αυτό βεβαίω είναι κυρίως στα χέρια των κρατών αλλά και των βουλευτών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σχόλια. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για την απάντηση στις ερωτήσεις αυτές. Το ερώτημά μου είναι θα μας τη στείλετε κιόλας. Γιατί έχουν πολλά και σημαντικά στοιχεία και εγώ θα τα ήθελα. Και τέλος, τέλος μία παρατήρηση από μένα. Η οδηγία περί αζωτούχων ε, είναι από τη δεκαετία του 1990, είναι πλέον πεπαλιωμένη και θα πρέπει να προσαρμοστεί στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στην κυκλική οικονομία και θα πρέπει ακριβώς να δούμε το τι αντιμετωπίζεται ως απόβλητο και θα πρέπει να δούμε ακριβώς την χρήση της ζωικής κοπριάς, η οποία εξακολουθεί ακόμα να υφίσταται διάκριση. Η και δεν τα έχει δει αυτά. Βλέπουμε λοιπόν πώς επηρεάζονται και οι οικογενικές επιχειρήσεις και τα ύδατα και το έδαφος. Ελπίζω λοιπόν να γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ναι. Δεν προγραμματίζουμε να γράψουμε και να δώσουμε γραπτό στις απαντήσεις αλλά θα ήθελα να αντιδράσω στο θέμα της οδηγίας, ε, το εάν είναι δηλαδή ε, απερχιωμένη ή όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι απερχιωμένη. Πρώτα απ' όλα γιατί καθορίζει στόχους, αφήνει στα κράτη-μέλη την επιλογή των αποτελεσματικότερων μέτρων και αυτό συνδυάζεται με το ότι τα σχέδια δράσης πρέπει να αναθεωρούνται κάθε 4 χρόνια. Οπότε η εφαρμογή της οδηγίας περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και τεχνολογικά στοιχεία. Επικαιροποιείται στην πράξη συνεχώς. Γι' αυτό τον λόγο η Κομισιόν δεν βλέπει τον λόγο αναθεώρησης της οδηγίας. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία των εδαφών και των υδάτων από τις γεωργικές πιέσεις και έχουμε ακριβώς και κάποια προσαρμοσμένα ειδικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα τεχνολογικά στοιχεία που αναπτύσσονται. Ευχαριστώ. Wij hebben ook de schriftelijke vragen ingediend Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το υποβάλαμε γραπτός. Ε, λάβαμε μια απάντηση. Αλλά θέλουμε να τα έχουν και οι συνεργάτες μας. Ε, εντάξει, δεν μπορούν να τα, να τα γράφουν τώρα, να κρατάνε σημειώσεις, στενογραφία και να τα γράψουμε εμείς. Αλλά θα θέλαμε να είναι διαθέσιμα από την Κομισιόν. Δηλαδή μας λέει ότι δεν μπορεί να στείλει τι απαντήσεις θα το ζητήσω μέσω της ομάδας μου, της ΕΛΚΑ, μέσω πιανού κανόνα, μπορούμε τελικά να τα λάβουμε μου φαίνεται περίεργο δηλαδή, πρέπει να σου το πω αυτό. Κυρία Πίρεκ, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να στείλει γραπτέ απαντήσεις. Και δεδομένε τις εμπειρίες που είχαμε με άλλε γενικέ διευθύνσει γνωρίζουμε ότι ακόμη και αν επιμείνουμε, δεν έχουν ε, κατά ανάγκη και τον έλεγχο. Οπότε δεν αλλάζει τίποτα. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να το σχολιάσετε κύριε Διευθυντά να προσθέσω ότι εφόσον λαμβάνουμε γραπτές ερωτήσεις υποβάλλουμε γραπτός και τις απαντήσεις. Αν στείλετε γραπτός τις ερωτήσεις πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσουμε γραπτός και εμείς. Κύριε Πρόεδρε, έθεσα γραπτές ερωτήσεις για την παρέκκληση. Ε, δεν έλαβα καμία απάντηση. Δύο γραπτές ερωτήσεις έχω δώσει και για τις προδιαγραφές. Καλώς. Ίσως το γραφείο σας μπορείτε, μπορεί να το λύσει διμερός με άλλους αρμόδιους διοικητικούς για να δούμε αν ήταν σωστή η μορφή της γραπτής ερώτησης, γιατί αν ήταν ε, η ενδεδειγμένη δεν βλέπω το λόγο για να έχετε λάβει απαντήσεις, ήταν εκτός της διαδικασίας. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή, ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση και ευχαριστούμε θερμά και τον Διευθυντή που ήρθε για να απαντήσει. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Αν δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα, η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 9 Ιουλίου στις Βρυξέλλες αυτή η συνεδρίαση.